Πιστεύουμε ότι και οι δύο πλευρέ, το Αρκτικό Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα υποφεληθούν από την συμμετοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση ω μόνιμο παρατηρητή στο Συμβούλιο. Γιατί θα, οι πολιτικέ μα και τα προγράμματά μα θα συντονιστούν καλύτερα εάν είμαστε παρόντε σε όλε τι δομέ του Αρκτικού Συμβουλίου. Οι γηγενεί πληθυσμοί είναι πολύ σημαντική εταίροι στην Αρκτική και θέλουμε να έχουμε έναν ευρύτατο διάλογο μαζί τους που θα βασίζεται σε μια ευρύτατη πολιτική υπέρ της υποστήριξης των γηγενών πληθυσμών που θα είναι επιτυχής και ούτως ή άλλως τη χρησιμοποιούμε και είναι και επιτυχής και σε άλλες χώρες του κόσμου. Η πρώτη προσπάθεια έγινε σε Βρυξέλλες το Μάρτιο. Θα ήθελα πολύ σύντομα να μιλήσω για τρεις τομείς όπου πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συνεισφέρει για να ενδυναμώσει τη διαχείριση του περιβάλλοντος στον Απότατο Βορρά μέσω της δουλειάς που κάνει κυρίως το Αρκτικό Συμβούλιο. Καταρχάς, το θέμα των κλιματικών δυνάμεων που αλλάζουν ε, το κάρβουνο, το μεθάνιο, που είναι παράγοντες που δεν παραμένουν πολύ στο περιβάλλον, αλλά που αλλάζουν ε, τα δεδομένα του κλίματος. Η κλιματική αλλαγή στην ε, ακτική ζώνη απαιτεί δράση και για αυτά τα αέρια σύντομης βραχίας διάρκειας, αλλά και για τα υπόλοιπα αέρια. Και υποστηρίζουμε τις ε, δράσεις του Ακτικού Συμβουλίου για να για να αντιμετωπίσει αυτά τα αέρια βραχία διάρκεια, εφόσον αυτό δεν μας αποτρέπει από την αντιμετώπιση και των υπολείπων αερίων. Καταρχάς, θα πρέπει να ασχοληθούμε με τα αέρια αυτά ε, και την μόλιση που προκαλούν στα πλαίσια το, της σύμβασης για τα αέρια ε, μεγάλου βεληνικούς ε, που μιλάει για όλα τα αέρια που μολύνουν το βόρειο ημισφαίριο και που είναι μια προσπάθεια που αντανακλάται και στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, η παρατήρηση και αξιολόγηση του προβλήματος, ούτως ώστε να καταλάβουμε καλύτερα τις περιβαλλοντικές τάσεις που υπάρχουν ε, στην περιοχή. Εδώ υπάρχει η πρωτοβουλία του, βιώσ... του παρατηρητηρίου για την Αρκτική, που... μια προσπάθεια που ξεκίνησε το Αρκτικό Συμβούλιο. Εμείς μπορούμε να συνεισφέρουμε στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ ε, των διαφόρων ε, δικτύων που υπάρχουν και των διαφόρων ε, εταίρων. Δεν θέλουμε να υπάρξει επικάλυψη προσπαθειών και θέλουμε τα κονδύλια να κατανεμηθούν πιο αποτελεσματικά. Η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος έχουν πολιτή εμπειρία και σε επίπεδο εταιρικής σχέσης, σε επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών, μέσω δικτύων κτλ και προσπαθούμε αυτή την εμπειρία να την χρησιμοποιήσουμε στα πλαίσια της, του παρατηρητηρίου αυτού για την Αρκτική. Το δεύτερο είναι μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Πριν τρία χρόνια υιοθετήσαμε την πολιτική αυτή και έκτοτε τα αποτέλεσματα της πολιτικής αυτής γίνονται ορατά σε όλη την Ευρώπη. Η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική βασίζεται στο γεγονός ότι είναι μοναδική αυτή η περιοχή και θα πρέπει να, αντιμετωπίσουμε, την αντιμετωπίσουμε με βιώσιμο τρόπο και να εμπλακούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Πιστεύουμε ότι η εμπειρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την ανάπτυξη μιας πραγματικά ε, ολοκληρωμένης ε, θαλάσσης πολιτικής μπορεί να βοηθήσει και την αρκτική ζώνη και την αρκτική, τις αρκτικές κοινότητες γενικά. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Ρέινολτς. Μπορούμε να αρχίσουμε την συζήτηση. Με την παρουσίαση της έκθεσης του εισηγητή μας, του κυρίου Γκάλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα προτιμούσα να σχολιάσω στο τέλος συνοπτικά, συνοψίζοντας. Αλλά ε, θα ήθελα να κάνω ορισμένες ερωτήσεις στους εμπειρογνώμονες. Καταρχήν σας ευχαριστώ για την επισκόπηση που παρουσιάσατε και για τις απόψεις σας για τις επιπτώσεις των κλιματολογικών αλλαγών όσον αφορά τις οδούς της ναυσιπλοείας και των τεκτενωμένων αυτή τη στιγμή από τα παράκτια κράτη τα οποία εφαρμόζουν συγκεκριμένες πολιτικές στα πλαίσια του Αρκτικού Συμβουλίου. Εάν έχουμε υπόψη μας αυτή την προοπτική, δηλαδή ότι ορισμένα πράγματα θα αλλάξουν κατόπιν των κλιματολογικών αλλαγών και θα ανοίξουν ε, οδοί ναυσιπλοείας νέοι, ε, θα επηρεαστεί και η προστασία του περιβάλλοντος στην περιοχή, αλλά ε, θα μπορέσει να υπάρξει και διερεύνηση για πετρέλαιο και αέριο στην περιοχή. Οπότε θα ήθελα να ρωτήσω τι, πώς θα επηρεάσει, ε, θα περάσουν αυτά τα στοιχεία τη διακυβέρνηση του χώρου. παρκούν οι νομικές διατάξεις, ε, οι, ε, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θαλάσσης ε, είναι κάτι που θα μπορέσει και στο μέλλον να καλύψει το θέμα ή θα χρειαστεί ένας, ένα νέο νομικό πλαίσιο. Εσείς ε, πιστεύετε ότι υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας ή ότι θα χρειαστούν ε, νέες νομικές συμφωνίες οι οποίες θα πρέπει να συναυθούν ιδίως πώς αξιολογείται το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στο χώρο. Είμαστε και εμείς νομοθέτες και η νομοθεσία μας ακόμη και αυτή τη στιγμή έχει έμεση επίπτωση στην περιοχή αυτή ακόμη και αν οι ίδιοι δεν έχουμε ε, μία παράκτια χώρα στην περιοχή. Πώς βλέπετε δηλαδή ότι θα υπηρεστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτές τις εξελίξεις. Ευχαριστώ κύριε Γκάλερ. Δίνουμε το λόγο. κύριο Γιάκον Τσάρη. Κυρία. Γιάκον για... που είναι σκιώδης εισηγήτρια από την ομάδα των συντηρητικών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε καθηγητά Γκερσόν, είπατε ότι δεν χρειαζόμαστε παροχημένες λύσεις. Θέλουμε ε, γρήγορες λύσεις που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ε, ανάγκες, αλλά που θα πρέπει να ληφθούν σχετικά γρήγορα για να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη μεταξύ των ενδιαφερομένων χωρών και να αποφευθεί κλιμάκωση των εδαφικών διεκδικήσεων και διαφορών. Η Αρκτική από μερικούς εκλεβάνεται ως το Ελντοράδο του Βορρά. Και γνωρίζουμε ότι οι πόροι βρίσκονται στο βόρειο τμήμα του πλανήτη, στο βόρειο ημισφαίριο, γι' αυτό όλοι σπέβδουν εκεί για να καρποθούν ένα τμήμα από το μερίδιο αυτών των φυσικών πόρων και του φυσικού πλούτου. Έχω μια ιδέα που δεν είναι δική μου προσωπική. Είναι ιδέα ενό γνωστού εξερευνητή του Βορρά. Το είπε και η Χίλαρη Κλίντον ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε για την αρκτική ζώνη ένα νέο μοντέλο διεθνούς συνεργασίας γιατί θα πρέπει βέβαια να ενισχύσουμε τη θέση του Αρκτικού Συμβουλίου, αλλά δεν έχουν πολύ εμπιστοσύνη σε αυτό το θεσμό. Σκέφτομαι λοιπόν, μήπως θα ήταν δυνατό και ζητώ τη δική σας ε, γνώμη, μήπως θα ήταν δυνατόν να συγκροτήσουμε μία επιστημονική διακλαδική μονάδα ομάδα μάλλον παρόμοια με αυτή που έχουμε για τις κλιματικές αλλαγές, ένα πάνελ εμπειρογνωμόνων που θα εξετάζει την κατάσταση στην αρκτική ζώνη και θα υποβάλει νομοθετικές προτάσεις ή προτάσεις για μέτρα που είναι κατάλληλα για την περιοχή ώστε να αποφύγουμε κλιμάκωση των εδαφικών διεκδικήσεων. Καλό θα ήταν να συσταθεί μια τέτοια ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων, επιστημόνων για την αρκτική αυτή ζώνη που θα συγκεντρώνει και πληροφορίες. Επίσης, καλό θα ήταν να υπάρχει ένα κέντρο πληροφοριών για την Αρκτική. Και μάλιστα ένα τέτοιο κέντρο υπάρχει στη Λαπωνία, που ήδη γιορτάζει την 20η επέτειο λειτουργίας του. Καλό, ήταν, καλό ήταν, λοιπόν να υπάρχει και ένα κέντρο πληροφόρηση για την Αρκτική. Θα συμβάλλει και αυτό στην διαμόρφωση και δραίωση εμπιστοσύνη μεταξύ των χωρών τη Αρκτική. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιάνστραμ για πέντε λεφτά. Κύριε Πρόεδρε, ήμουν μέλος της τοπικής κυβέρνησης ε, του Αμβούργου και πάντοτε ασχοληθήκαμε με το λιμάνι του Αμβούργου που είναι το μεγαλύτερο λιμάνι στην περιοχή και το δεύτερο μεγαλύτερο στην Ευρώπη και ε, πριν λίγο η εταιρεία Μπελούγκα προσπάθησε να δει αν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη διέλευση ε, από βορρά προς την Ασία. Ε, τι χρειάζεται ε, για να γίνει αξιόπιστη αυτή η εναλλακτική λύση και πώς πιστεύετε ότι θα αναπτύξει μακροπρόθεσμα η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη διέλευση η οποία είναι πολύ σημαντική ε, και ποιος είναι ο ρόλος, ποιες είναι οι δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στις διάφορες συνελεύσεις οι οποίες ασχολούνται με τα θέματα της της Αρκτικής. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Λέτζινγκ, η οποία είναι σκιώδη συγγήτρια για την ΚΟΕ, για την Ενωμένη Αριστερά. Μικρόφωνο παρακαλώ. Τώρα με ακούτε καλύτερα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και πάλι για τις σημαντικές πληροφορίες διότι ασχολούμαστε και πάλι αυτό το θέμα το οποίο θα έχει μεγάλη σημασία στο μέλλον. Έχω διαβάσει πάρα πολλές αναλύσεις όπου ορισμένα αντικρούν αυτά τα οποία μας είπε ο κύριος Ιμιούνατσον. Δηλαδή διαβλέπονται πολλές διαμάχες στο μέλλον μέλλον και ότι θα υπάρχουν γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις στο μέλλον. Πιστεύω ότι αυτή είναι μια μεγάλη πρόκληση για την επίλυση πολιτικών διαμαχών και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παίξει ένα θετικό ρόλο σε αυτό το θέμα. Όσον αφορά την καταστροφή στον κόλπο του Μεξικού, το ΒΒΕΦ και άλλες διεθνείς οργανώσεις όσοι ζητούν να υπάρξει ένα μορατόριουμ σχετικά με την ανάπτυξη της εξορίξεως πετρελαίου στην Αρκτική. Τι σκέφτεστε γι' αυτό και κύριε Γκάλερ θα ήθελα να σας ρωτήσω και εσάς πιστεύετε ότι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο επαρχεί τι θα μπορούσε κανείς να κάνει και μήπως θα έπρεπε να βασιστούμε εις το πρόγραμμα σαν πρότυπο. Μήπως ε, πιστεύετε ότι χρειαζόμαστε ένα νομικό οικοδόμημα σαν την ε, Συμφωνία Άρκτικ όπου η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξετάζει διάφορα θέματα όπως και την εκμετάλλευση του πετρελαίου διότι εδώ και πολλά χρόνια οι παράκτες χώρες από απορρίπτουν αυτή τη συμφωνία και αναρωτιέμαι αν δεν θα ήταν η καλύτερη λύση για να μπορέσουμε να αποδυναμώσουμε ε, τις διαμάχες και ε, να δημιουργήσουμε μία αποστρατικοποιημένη περιοχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Κόβαλ, πέντε λεφτά. Ευχαριστώ. Ε, η ομιλία του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας έδωσε πληροφορίες για την αρκτική ζώνη και μας μίλησε για μία συνάντηση που είχε με εκπροσώπους των αρκτικών χωρών. Έχω δύο ερωτήσεις. Ποιες είναι οι διατάξεις ε, που ισχύουν σε ό,τι αφορά τις ε, ενώσεις για τον πληθυσμό της Αρκτικής. Γιατί μας έδωσε κάποια στοιχεία τέτοιων ε, συζητήσεων που γίνονται μεταξύ των ε, γηγενών πληθυσμών. Επίσης, θέλω να δω ποια είναι η θέση μας απέναντι στη θέση αυτών των γηγενών πληθυσμών. Τους αντιμετωπίζουμε με τον δέοντα σεβασμό Επίσης αυτοί, α, αυτοί οι πληθυσμοί, οι γενείς πληθυσμοί, αλλά και κάποιες εθνοτικές κοινότητες έχουν και δικά τους κράτη. Δεν είναι μόνο οι δικές μας ευρωπαϊκές αρκτικές χώρες, αλλά και οι μεταξύ τους σχέσεις. Ποιες είναι μεταξύ των αρκτικών χωρών, αλλά και των αρκτικών εθνών. Ποιες είναι οι σχέσεις μεταξύ τους και ποιες είναι, και ποιες είναι και οι απόψεις και οι θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά τι σχέσει μεταξύ των διαφόρων εθνοτήτων και κρατών τη Αρκτική. Ευχαριστώ. Για την Μάκη. Σκιώδης εισηγήτρια των φιλελεύθερων για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή τον κύριο Γκάλερ που διοργάνωσε αυτή την ακρόαση και τη συζήτηση που κάνουμε για την αρκτική ζώνη. Είναι πολύ καλό που το κάνουμε αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται το Κοινοβούλιο να δραστηριοποιηθεί και να συμμετάσχει στις συζητήσεις να... και να προωθήσει πρωτοβουλίες. Επίσης, καλό να τονιστεί ο ρόλος του φαινομένου του θερμοκηπίου και της κλιματικής αλλαγής ε, και πώς επηρεάζει το περιβάλλον στην Αρκτική. Θα πρέπει να κάνουμε μελέτες ε, επιπτώσεων στο περιβάλλον. Επίσης, ένα δεύτερο θέμα είναι τα δικαιώματα των ε, γηγενών πληθυσμών. οι Σάμοι που είναι παρόντες στην ε, Λαπωνία και οι υπόλοιποι γηγενείς πληθυσμοί, ε, το μόνο εργαλείο που έχουν είναι να εκφράσουν τη γνώμη τους. Και εμείς πρέπει να πω και τα ακτικά κράτη αλλά και εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε δράσει με παραδειγματικό τρόπο. Πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος μεταξύ των ΣΑΜΙ, του Κοινοβουλίου και των κρατών μελών. Δεν μπορούν να ληφθούν πολιτικές αποφάσεις χωρίς ε, να ακούσουμε τους λαούς αυτούς για τους οποίους ε, προωθούμε αυτές τις πολιτικές. Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας για τον τακτικό διάλογο και τη σημασία του. Τι διευθετήσεις ετοιμάζονται για να δημιουργηθεί αυτός ο, ο διάβλος ε, μόνιμης επικοινωνίας. Η Λίζα Γιάκοψον από τα αριστερά μίλησε πολύ σοφά. Κυρία Γιακονσάρη. Θα πρέπει να υπάρξει ένα κέντρο ενημερωτικό για την Αρκτική ή μάλλον υπάρχει στο Ρωμανιάμι. Καλά είναι αυτά που μας είπε, γιατί ένα τέτοιο κέντρο ε, εξυπηρετεί, θα εξυπηρετήσει και το αρκτικό δίκτυο. που είναι διεθνές δίκτυο. Και νομίζω ότι μπορεί να προωθήσει συνεργασία σε διάφορα επίπεδα. Ευχαριστώ τον κύριο Γιατενμάκη. Θα πρέπει να σας μειώσω το χρόνο κατά το ίμιση στους επόμενους ομιλητές. Γιατί βλέπω ότι μακραίνει ο κατάλογος και μην ξεχνάμε ότι ο εισηγητής και 10.30 θα πρέπει να μας εγκαταλείψει. Μετά λοιπόν τους εισηγητές θα πρέπει να μιλήσει και εκείνος. Ε, Επομένω, έχετε το μισό χρόνο, δυόμιση λεπτά. Κύριε Πρόντι, δυόμιση λεπτά λοιπόν κι εσεί. Είναι πολύ σημαντική αυτή η ακρόαση, Πρόεδρε. Κυρίως γιατί πρέπει να προβληματιστούμε για τους φυσικούς πόρους. Αυτή τη στιγμή η Ρωσική Ομοσπονδία με τον Πούτιν έστησε την σημαία της στο Βόρειο Πόλο ε, μάρκαρε ουσιαστικά την περιοχή της όπως κάνουν τα ζώα. Θεώρησε ότι είναι εθνικό έδαφος. Και επομένω θεωρεί ότι έχει και άμεση πρόσβαση στους φυσικούς πόρους. Πρέπει να σκεφτούμε το θέμα αυτό όχι μόνο για την αρκτική περιοχή, αλλά επειδή για την αρκτική περιοχή ξεκινάμε πραγματικά από το μηδέν. Ε, ίσως λοιπόν θα ήταν ένα καλό φυτόριο η αρκτική. Ε, να ξεκινήσουμε από την υπόθεση ότι οι φυσικοί πόροι είναι περιορισμένοι και επομένως επειδή υπάρχει μια άλλη εξάρτηση όλες οι χώρες εξαρτώνται από αυτούς τους ε, περιορισμένους φυσικούς πόρους, θα πρέπει να κάνουμε μια συνενετική διαχείριση των πόρων, μια και δεν είναι περιόριστες, Αν ακριβώς θέλουμε να αποφύγουμε συγκρούσεις και σειράξεις. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε με πειραματικό τρόπο από την αρκτική ζώνη για να δούμε ε, αν μπορούμε, να δούμε αν μπορούμε να προωθήσουμε την πολιτική και όχι τη βία. Θα ήθελα και εγώ να σας μιλήσω για τους γηγενείς πληθυσμούς. Το Μάιο συμμετείχα στη συνεδρίαση που, που έκαναμε για να μιλήσουν οι γηγενείς πληθυσμοί για τη θέση τους και για τα δικαιώματά τους. Ακόμη και εδώ η Αρκτική θα μπορούσε να είναι ένα εργαστήρι για να πειραματιστούμε για το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μηχανισμούς απόφασης, συνενετικούς και πώς μπορούμε να επιδιορθώσουμε αυτή τη θέση ληστείας την αρπακτική θέση που είχαμε απέναντι σε αυτούς τους λαούς, ε, σφετεριζόμενοι τα δικαιώματά τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έρχομαι από μία από αυτές τις χώρες οι, οποίες ε, είναι, η οποία είναι παράκτια της Αρκτικής, από τη Δανία, ε, από τη Γρυλανδία. Αλλά η Γρυλανδία εσκεμμένος ε, Ρίψε ε, την συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Γρυλανδία βρέθη ε, προσφάτως πετρέλαιο. Βλέπουμε όμως τώρα ότι οι κάτοικοι της Γρυλανδίας στρέφονται μάλλον προς την Αμερική από ότι προς την Ευρώπη. Μόνο τρεις ε, χώρες ε, ε, πλήττονται από περιέχονται στις παράκτες της Ακτικής και όχι η Σουηδία και η Νορβηγία. Είμαι μέρος της αντιπροσωπείας με τον Καναδά και ρώτησα τι γίνεται με τη διέλευση την βορειοδυτική και τι θα έπρεπε κανείς να πληρώνει σαν για να περάσει ε, και με δισταγμό μου απάντησαν μάλλον θα μπορούσα να σας πω ότι ουσιαστικά δεν μου απάντησαν είναι ένα θέμα που θα πρέπει να συζητηθεί αλλά δεν βλέπω σαν Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε τη δυνατότητα να επηρεάσουμε ε, ουσιαστικά την κατάσταση. Ευχαριστώ δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ. Η συζήτηση αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα και εγώ είμαι υπέρ μια συντονισμένη πολιτική για την αρκτική ζώνη και θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε, γιατί νομίζω ότι οι εταίροι μας επιτάχυναν τις ενέργειες και δραστηριότητες τους στην περιοχή. Έχω μια ερώτηση προς τους δύο καθηγητές. Μήπως υπάρχει κάποια μελέτη ή έχετε γνώμη σε ό,τι αφορά την αύξηση των μεταφορών στην αρκτική ζώνη, στον αρκτικό κύκλο. Πιστεύετε ότι εξαιτία τη αύξηση των μεταφορών θα επιταχυνθεί το λιώσιμο των πάγων στον αρκτικό κύκλο. Κάτω από τον πάγο υπάρχουν νησιά που δεν ανήκουν σε καμία χώρα. Και τι θα γίνει αν λιώσουν οι πάγοι πάνω από τα νησιά αυτά με τις κλιματικές αλλαγές δυόμιση λεπτά προς τον κύριο Τάνοκ. Ευχαριστώ. Ε, οι περισσότερες ερωτήσεις που ήθελα να θέσω ετέθησαν την κυρία Ρόσμπακ. Με σε ενδιέφερε το καθεστώς της Γκρινλάκ, της ε, συγγνώμη. Η εξωτερική τους πολιτική ασκείται από την κυβέρνηση της Δανίας και είναι εξαρτώμενο έδαφος, το οποίο όμως έχει μία τάση προς την ανεξαρτησία. Ε, δεν νομίζω ότι, ο τρόπος αυτός να ασκείται η εξωτερική πολιτική της Γρυλανδίας από το Υπουργείο Εξωτερικών της, της Δανίας δεν είναι ο καλύτερος τρόπος. Κάποιος από την ΚΟΕ νομίζω είπε ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε τους φυσικούς πόρους στην Αρκτική. Γιατί να διατηρήσουμε πράγματα ε, κάτω από την ε, επιφάνεια της θάλασσας ε, που υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια όπως πετρέλαιο και φυσικό αέριο Νομίζω ότι είναι ανόητη αυτή η ιδέα ότι είναι, ανήκουν στη φύση ας πούμε και ότι δεν πρέπει να τα αγγίξουμε. Φυσικά θα πρέπει να σεβαστούμε το δίκαιο και να υπάρξει μια συνεργασία. Ε, νομίζω, δεν ξέρω αν μπορούμε να συγκρίνουμε την Αρκτική με την Ανταρκτική. Δεν νομίζω. Αλλά η ιδέα ότι πρέπει να σταματήσουμε τις εξορίξεις ε, πετρελαίου και φυσικού αερίου από το βυθό της θάλασσας δεν ε, είναι γελία. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο στους Καναδούς, στους Αμερικανούς και στους Ρώσους να σταματήσουν ε, τις προσπάθειες αυτές τη στιγμή που υπάρχει ανάγκη, υπάρχουν τρομακτικές ενεργειακές ανάγκες. Ευχαριστώ τον κύριο Τάνοκ. Τώρα θα δώσω το λόγο στους εμπειρογνώμονες. Θα ξαναμιλήσουμε τη σειρά με την οποία έκανα τις παρουσιάσεις τους, τις αρχικές. Το πολύ πέντε λεφτά ο καθένας, σας παρακαλώ. Και κανονίστε μεταξύ σας ε, ποια ερώτηση σας αφορά, να την απαντήσετε. Ε, ο κύριος, ο καθηγητής Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να απαντήσω σε δύο ερωτήσεις τουλάχιστον. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά αυτή, αυτόν τον αγώνα για την αξιοποίηση των πόρων, την κούρσα, ποιος θα πρώτο ε, εκμεταλλευτεί αυτούς τους πόρους της Αρκτικής. Νομίζω ότι έγινε μια παρανόηση εδώ και ο λόγος αυτής της παρανόησης οφείλεται στο ότι, κατά τη γνώμη μου, η ορολογία κούρσα για τους σπόρους προϋποθέτει ανταγωνιστές που ξεκινούν έναν αγώνα, μια κούρσα για πόρους που δεν ανήκουν σε κανένα και δεν είχαν αξιοποιηθεί μέχρι στιγμής. Η ε, πόροι που βρίσκονται όμως ε, στο έδαφος μιας ε, χώρας είναι ιδιοκτησία αυτή της χώρας. Δεν υπάρχει θέμα κούρσας ή ανταγωνισμού μεταξύ διαφόρων χωρών. Όσοι βρίσκονται ε, στη γη των ε, ε χωρών είναι δική τους ε, ιδιοκτησία, ανήκουν στη δική τους κυριότητα με βάση εθνική και διεθνή νομοθεσία. Οπότε αυτή η ορολογία ο αγώνας ή η κούρσα για τους ε, φυσικούς πόρους δεν είναι σωστή, δεν είναι δόκιμη για την Αρκτική. Γιατί υπάρχουν οι πόροι, αλλά ανήκουν ήδη στις ε, συγκεκριμένες αρκτικές χώρες. Δεν είναι αδέσποτη αυτή η φυσική πόρη της Αρκτικής. Τώρα, σε ό,τι αφορά το καθεστώς διακυβέρνηση, αν είναι επαρκές, αν χρειαζόμαστε περαιτέρω διεθνείς ε, διατάξεις και κανονισμούς, και επίση υπάρχει και συζήτηση για το κατά πόσο χρειαζόμαστε μια συνθήκη για την Αρκτική. Γιατί έχει πολλές ιδιαιτερότητες ο αρκτικός κύκλος και ίσως ε, διαφέρει από αυτά που ισχύουν για το διεθνέ δίκαιο των ωκεανών. Όλοι συμφωνούν για την ιδιαιτερότητα του αρκτικού κύκλου και πιστεύω ότι ο αρκτικό ωκεανός είναι ιδιάζων γιατί έχει θαλάσσιο πάγο και για το θαλάσσιο πάγο δεν ισχύει διεθνές δίκαιο. Η συνθήκη για τις θάλασσες ε, του 1982 απαρτίζεται από 320 διαφορετικά άρθρα. Τα άρθρα 1, 2, 3 και 4 αφορούν τα ε, ύδατα στα οποία υπάρχει πάγος, αλλά δεν υπάρχει ειδικό δίκαιο για το θαλάσσιο πάγο. Δηλαδή, αυτός ο πάγος των θαλασσών θεωρείται έδαφος γιατί μπορούν ακόμη και αεροπλάνα να προσγειωθούν σε πάγο ή υπάρχουν πάγοι που ε, παρε, παρε, στους ωκεανούς ε, κυκλοφορούν, μετακινούνται κατά κάποιο τρόπο δηλαδή είναι έδαφος αλλά υπό κάποια έννοια είναι και είδωρ και εξυπηρετεί και τους ε, δύο σκόπους και λειτουργίες. Για πολλά χρόνια στην ακτή δεν μπορούσαν να περάσουν ε, πλοία. Σήμερα όμως περνάνε πλοία από πολλές περιοχές της Αρκτικής. Οπότε είναι πλωτή θάλασσα σε μεγάλο ε, βαθμό η Αρκτική με βάση είναι ανοιχτή θάλασσα με βάση την τρίτη συνθήκη για την ανοιχτή θάλασσα. Άλλο, άλλη μορφή είχε ο θαλάσσιος πάγος στη δεκαετία του 60 και του 70 και άλλη μορφή έχει σήμερα. Επίσης, κάποιες διατάξεις εφαρμόθηκαν από τον Καναδά και τη Ρωσία, αλλά και γίνονται συζητήσεις ε, και στον Καναδά και στη Ρωσία για το κατά πόσο ο θαλάσσιος πάγος θα πρέπει να θεωρηθεί ως έδαφος. Δηλαδή, τι εστί θαλάσσιος πάγος και μπορεί να δημιουργήσει πρόσφορα έδαφος για συγκρούσεις αυτή η έννοια του πάγου των θαλασσών. Ευχαριστώ. και Μούντρασον. Για να απαντήσει ο ίδιος. Όχι πάνω από πέντε λεφτά παρακαλώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα ενδιαφέροντα σχόλιά σας. Θα ήθελα να απαντήσω σε διάφορα σημεία. Σε ό,τι αφορά τα υπάρχοντα πλαίσια και τις ε, συμβάσεις. Ε, το δίκαιο της θάλασσας του ΟΗΕ είναι το βασικό α, διεθνές πλαίσιο για την Αρκτική. Όπως ανέφερα όμως και στην παρουσίασή μου, Υπάρχει μια αμφισημία. Θα πρέπει να στραφούμε προς το 2013 και 2014 ε, γιατί η Δανία θα διεκδικήσει εξ ονόματος της Γρυλανδίας ε, θα κάνει δηλαδή τις εδαφικές της ε, διεκδικήσεις. Και ο Καναδάς επίσης που υπέβαλε τις αρχικές του διεκδικήσεις το 2001 θα τις επαναδιατυπώσει. οι Καναδοί και οι Δανείοι, ας πούμε, ε, έχουν διαφορετικές αποσιωσμένα θέματα από τους Ρώσους. Επίσης, η ρητορία η υπεριαλιστική ρητορία του 19ου αιώνα ε, έχει κάποιες αναλογίες με, το τι, με τη ρητορία για την Αρκτική. Για τη Γρυλανδία. Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Τι θα συμβεί με τη Γρυλανδία και ποια είναι η θέση της. Γιατί αυτό συνδέεται και με, την, με το καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δανία, Σουηδία και Φιλανδία. Ε, έχουμε τρία ευρωπαϊκά κράτη τα οποία είναι τέρη, ενώ η Γρυλανδία δεν είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Γρυλανδία και η Σουηδία δεν έχουν ακτογραμμή στην Αρκτική. Όταν συναντούνται αυτά τα πέντε κράτη, υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα επίσης και με το καθεστώς του παρατηρητή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Αρκτικό Συμβούλιο. Οι Ρώσοι, Φερρυπίν, θεωρούν ότι όσοι λιγότεροι στο Αρκτικό Συμβούλιο τόσο καλύτερα. Δεν θέλουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κίνα και τον ΝΑΤΟ να μπουν στην περιοχή. Να το πούμε και αυτό είναι ενδιαφέρον. Πολύ τονίσατε πολύ σωστά τα δικαιώματα των γηγενών πληθυσμών και πρέπει να πούμε ότι η επιρροή τους αυξάνεται. Καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούν να αποκλειστούν. Είναι εταίροι και αυτοί, είναι εμπλεκόμενοι, ενδιαφερόμενοι και όσο περισσότεροι οι ενδιαφερόμενοι και οι εμπλεκόμενοι, τόσο μεγαλύτερη συζήτηση για τη διακυβέρνηση. Ε, στη συνάντηση του Καναδά, ε, ο αποκλεισμός των ε, υπολείπων αρκτικών κρατών δεν έγινε δεκτός με καλό τρόπο. Για τα τεχνικά θέματα δυστυχώς δεν είμαι εμπειρογνώμονας. Μπορώ να απαντήσω λίγο πρώτος ομιλητής μετά για τα τεχνικά θέματα. Και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια και μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω την, ε, της διεθνούς συνεργασίας και της διασυνοριακής, των διασυνοριακών ε, διαδικασιών, παίζει ένα ρόλο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή ενδιαφέρεται για το εμπόριο, έχει ε, αντίστοιχη στάση με, την, με τη ΣΥΠΑ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρότι δεν έχει άμεση πρόσβαση αυτή τη στιγμή και δεν είναι μέλος του Αρκτικού Συμβουλίου ακόμα τουλάχιστον, δεν μπορεί να αποκλειστεί μακροπρόθεσμα. Και η Κίνα το ίδιο. Και η Ιαπωνία. Θα εισβάλλουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ε, στη, τελικά οι μεγάλοι αυτοί εταίροι. Γι' αυτό λοιπόν καλό θα ήταν να υπάρχει ένας μηχανισμός να ακουστούν οι απόψεις σε υψηλό επίπεδο όλων. Ευχαριστώ τον ε, καθηγητή Ίγκη Μούντερσον και τώρα ο κύριος Ρέινολτς από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Δυστυχώς θα πρέπει να σας δώσω μόνο τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος. Καταρχήν όσον αφορά τη διακυβέρνηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η, ε, θεωρεί ότι θεωρούμε σαν σημείο αναφοράς τη θέση η οποία πρεσβεύεται στην ανακοίνωση του 2008 δηλαδή ε, να βασιστούμε στο UNCLOS, στη σύμβαση UNCLOS και να εφαρμόσουμε τις ισχύουσες υποχρεώσεις αντί για νέα νομοθετικά μέσα. Πράγμα που δεν αποκλεί να αναπτύξουμε τις συμφωνίες ή να καλύψουμε με νέες συμφωνίες τα κενά που ενδέχεται να υπάρχουν ε, συγκεκριμένα στο περιβάλλον. Συμφωνώ ότι η Ανταρκτική αυτή τη στιγμή δεν συζητείται και ιδίως διότι ε, δεν ε, ε, στηρίζεται από τα κράτη της Ανταρκτικής και λόγω των σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ των κρατών της Αρκτικής και της Ανταρκτικής και που αναφέρθηκαν. Όσον αφορά την αξιολόγηση των πληροφοριών, αν δηλαδή θα έπρεπε να έχουμε κάτι σχετικό με το, ε, ε, τη στρογγυλή τράπεζα για την Αρκτική και στην Ανταρκτική. Πιστεύουμε ότι ήδη υπάρχει μια επαρκής υποδομή ε, συνεργασίας όσον αφορά την έρευνα, την αξιολόγηση ιδίω όσον αφορά την Αρκτική και πιστεύω ότι θα πρέπει να συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια και θα θέλαμε να δούμε πώς αυτό μπορεί να λειτουργήσει προτού εξετάσουμε νέες δομές οι οποίες θα δημιουργήσουν ορισμένες επικαλύψεις. Το Κέντρο Πληροφοριών της Αρκτικής αναφέρθηκε, συζητείται το θέμα. Θα έχουμε εξελίξεις και κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα ε, ενδιαφέρουσες. Πολλοί αναφέρθηκαν στους ηθαγενείς. Τι θέλουν, τι μπορεί να κάνει για αυτούς η Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι ορισμένες απαντήσεις έχουν δοθεί διότι Ε, ένας παρεμβαίνων είπε ότι ουσιαστικά πρέπει να βελτιώσουμε τις δυνατότητες διαλόγου και να ακούσουμε πλέον προσεκτικά τα, τους ηθαγενείς να εξασφαλίσουμε ότι οι θέσεις τους ε, συμπεριλαμβάνονται στις ε, νομοθετικές προσπάθειες Ευρωπαϊκής Ενώσεως και αναφέρουμε εδώ στον συγκεκριμένο ρόλο της ε, κοινότητας της Αρκτικής που έχουν ειδική θέση εις ε, τα θεσμικά όργανα της περιοχής και πρέπει να το σεβαστούμε. Δεν νομίζω ότι απάντησα σε όλα τα σημεία αλλά νομίζω τα υπόλοιπα μπορώ να τα αφήσω τα τελικά σχόλια από την ε, κυρία Γκάλερ, από τον κύριο Γκάλερ, συγγνώμη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους συζητητές που παρουσίασαν το θέμα και νομίζω ότι στη συζήτηση ορισμένα θέματα διευκρινίστηκαν και καθορίστηκαν γραμμές τις οποίες πρέπει να ακολουθήσουμε στην περαιτέρω δράση μας. Βέβαια ο, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μέτοχος στην αλλά έχουμε συγκεκριμένα συμφέροντα είμαστε παρόντες με τα προγράμματά μας με το πρόγραμμα πλαίσιο ερεύνης με τους κανόνες ναυτιπλοείας για την εμπορική ναυτιλία και για τον αλληλευτικό στόλο και έχουμε και συγκεκριμένη νομοθεσία μας ενδιαφέρει η Αρκτική αναφερθήκαμε στις κλιματολογικές αλλαγές που πλήττουν την Αρκτική περιοχή πιο γρήγορα από ό,τι αλλού και είναι και πιο προφανείς οι αλλαγές αυτές ε, υπάρχει μία πτυχή προστασίας περιβάλλοντος στο θέμα αυτό είναι δηλαδή ένα θέμα το οποίο πρέπει να ενδιαφέρει όλους και την Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό θα ήθελα να αναφέρω ότι θα συζητηθεί το θέμα ε, του περιβάλλοντος με τη Ζακλίν Μακλέιτ της ε, Ευρωπαϊκής, ε, του Ευρωπαϊκού Γραφείου Περιβάλλοντος που δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα αλλά θα έρθει για πρωινό στις 15 Σεπτεμβρίου και θα εμβαθύνουμε περισσότερο το θέμα αυτό. Επίσης ε, αναφερθήκαμε και στους Ιθαγενείς, οι Σάμι στην Ευρώπη, οι Νουίτ στον Καναδά και στις Ηνωμένε Πολιτείες η προστασία του περιβάλλοντος και τα δικά του συμφέροντα των ηθαγενών αυτών δηλαδή ε, ε, συμβαδίζουν και πρέπει να καλυφθούν οι απαιτήσει τους για μία βιώσιμη ανάπτυξη και όχι διατήρηση διότι άκουσα ότι ορισμένοι ε, λέγουν δεν ζω σε ένα μουσείο δεν θέλω να μείνουν τα πράγματα ως έχουν πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη στην περιοχή μου και πιστεύω ότι αυτό ισχύει και για τους ηθαγενείς αλλά και για αυτούς οι οποίοι διαβιούν εκεί χωρίς να είναι ηθαγενείς. Δεν πρόκειται για μεγάλους πληθυσμούς και ε, υπάρχει επίσης το θέμα των εκμεταλλεύσεων των πρώτων υλών μας ενδιαφέρει ε, το πετρέλαιο και το αέριο αλλά έχουμε σοβαρές προδιαγραφές και οι βόρειοι εταίροι μας οι Ισλανδοί και οι Νορβηγοί έχουν ε, αυστηρές προδιαγραφές για το περιβάλλον μπορούμε να συνεργαστούμε στενά και καλά και να σε σαν τη Ρωσία που δεν χρησιμοποιεί αυτές τις προδιαγραφές ενδέχεται να μπορέσει να συνεργαστεί ε, και να εξασφαλίσει ότι θα χρησιμοποιήσουμε υψηλές προδιαγραφές ε, κατά την ε, εκμετάλλευση αυτού του χώρου της Αρκτικής. Είμαι πεπισμένος ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να έχει έναν μόνιμο παρατηρητή στο Αρκτικό Συμβούλιο και για τα κράτη οι μελη που έχουν, βρίσκονται μακριά από την Ακτική θα έπρεπε να έχουμε έναν εκπρόσωπο μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Αρκτικό Συμβούλιο διότι μπορούμε έτσι να ενημερωνόμαστε για τα θέματα της ναυτιλίας, του περιβάλλοντος, της έρευνας αντί να έχουμε μεμονωμένα κράτη ε, τα οποία έχουν αναθέσει ορισμένες αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όπου θα έπρεπε να μπορεί να ε, εκπροσωπείται τουλάχιστον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η, ε, η Αρκτική είναι είτε εδαφικά ύδατα είτε ε, διεθνή ύδατα τα οποία δεν ε, ελέγχονται από κανένα κράτος και γι' αυτό θα έπρεπε ε, να υπερισχύσει η συμφωνία άρκτης ε, άλλων ενδεχομένων και ε, τέλος πρέπει να πω ότι όλοι ενδιαφερόμαστε να μην υπάρξει σταρατικοποίηση για οποιοδήποτε λόγο δεν υπήρξε κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου και από το τέλος του ψυχρού πολέμου επίσης και στο μέλλον νομίζω ότι δεν θα πρέπει να υπάρξουν μόνιμες στρατιωτικές εγκαταστάσεις ή ε, άλλες ε, ε, τέτοιες εγκαταστάσεις στο μέλλον. Σας ευχαριστώ όλους. Φαντάζομαι ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε το διάλογο και σαν εισηγητής είμαι στη διάθεσή σας για να συνεργαστώ με τους κοιόδης εισηγητές και όποιος συνάδελφος θέλει να παρέμβει είναι ευπρόσδεκτος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γκάλερ. Ευχαριστώ και τους φιλοξενούμενους μας, ε, τους ε, εμπειρογνώμονες. Από τις 13 έως τις 15 Σεπτεμβρίου μου είπαν ότι θα γίνει μία διάσκεψη του Κοινοβουλίου για την Αρκτική Ζώνη. Όσοι ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε μπορείτε να γράψετε το όνομά σας και να σημειώσετε ότι θα λάβει χώρα αυτή τη διάσκεψη. Για την έκθεση Γκάλερ θέλω να πω ότι θα παρουσιαστεί στην επόμενη, σε μία από τις επόμενες 26 και 27 Οκτωβρίου. Πάμε στην επόμενη, στο επόμενο σημείο της Μεσίας Διάταξης, πρόταση ψηφίσματος. Hepkins. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω κατάχρηση της καλοσύνης σας και να θέσω ένα ζήτημα με ερωτηματικό στο τέλος γιατί δεν είμαι βέβαιος. Ο κύριος ε, Σέρς που όπως ξέρετε έχει στενές σχέσεις με το Πακιστάν οργάνωσε μια συνεδρίαση χθε και μάλιστα παρότεινε τους συναδέλφους να ασχοληθούν και να διαφερθούν για τις πλημμύρες στο Πακιστάν εν ώψη της, του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών την επόμενη εβδομάδα που θα ασχοληθεί και με το σημείο αυτό. Και μάλιστα μου ζήτησε επειδή είμαι μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων να επιστήσω την προσοχή σας στην κατεπίγουσα κατάσταση του Πακιστάν και στην ανάγκη να αναλυφθεί επιγόντως δράση. Διαρωτώ με λοιπόν κύριε Πρόεδρε, μήπως θα μπορούσαμε να βρούμε κάποιο τρόπο στο εγγύς μέλλον κατά προτίμηση ίσως ε, σε μια έκτακτη συνεδρία στη Δευτέρα στο Στρασβούργο για να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Γιατί συνάδελφοι από όλες τις πολιτικές ομάδες ενδιαφέρονται για το ζήτημα αυτό. Και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε την ανάμειξη και την παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο θέμα των πλημμυρών του Πακιστάν. Πολύ ωραία. Δέχομαι την πρόσκλησή σας. Και θα κάνω ό,τι μπορώ, ούτως ώστε να τεθεί το σημείο αυτό στη μερίσια διάταξη της ε, Επιτροπής μας. Ξέρετε όμως ότι στην Ολομέλεια, την επόμενη, προβλέπεται μια συζήτηση για το θέμα αυτό. Και στη συνεδρίαση για την ανάπτυξη που αφορά κυρίως τις ανθρωπιστικές βοήθειες, εκεί έχει ενταχθεί αυτό το σημείο. Φυσικά η πρότασή σας ε, είναι απόλυτα αποδεκτή και μετά από την ε, συζήτηση που θα γίνει στα πλαίσια τη Ολομέλεια για την Ανάπτυξη, κάπου θα, θα το ξαναβάλουμε και στη συνεδρίαση τη δική μα Επιτροπή. Το σημείο 2. Πρόταση ψηφίσματο για την ενίσχυση τη ΟΑΣΕ και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωση. Έχουμε ήδη συζητήσει αυτό το σημείο στις 22 Ιουνίου στην Ολομέλεια για την ευρωατλαντική αρχιτεκτονική δομή για θέματα ασφάλειας και στα πλαίσια αυτά συζητήσαμε για την ΟΑΣΕ. Από την υιοθέτηση της τελικής πράξης του Ελσίνκη, η οργάνωση για την ασφάλεια και την συνεργασία στην Ευρώπη ε, έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην δομή της ευρωατλαντικής και ευρωατλαντικής ασφάλειας. Το 1999 ε, ήταν η τελευταία μεταρρύθμιση της ΟΑΣΕ μετά από το δύο χρόνια συζήτηση που έγιναν ε, στα πλαίσια της διαδικασίας ε, της, του, της Κέρκυρας. Και ο πρόεδρος ο τότε ε, συγκάλεσε μια νέα σύνοδο για την ΟΑΣΕ το Δεκέμβριο με σκοπό να αναπτυχθούν μηχανισμοί πιο ευέλικτοι και να δοθεί μια νέα όθηση και μια νέα αξιοπιστία στη δραστηριότητα αυτής της οργάνωσης. Θα θέλαμε λοιπόν να συμμετάσχουμε και εμείς αυτή τη συζήτηση, γιατί η Ένωση ε, παίζει το ρόλο της ε, στη Σύνοδο Κορυφής. Πρέπει να παίξει το ρόλο στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου ούτω ώστε να διατρανωθεί η σημασία αυτή τη σημαντική κατά διεθνού οργάνωση. Ο κύριος Ράουτσεκ θα ήθελα να μας παρουσιάσει τις βασικές πτυχές του κειμένου του ψηφίσματός του. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως είπατε ήδη, η ΟΑΣΕ έγινε τμήμα της αρχιτεκτονικής δομής ε, της ε, ευρωατλαντικής και ευρωασιατικής ασφάλειας. Ε, είναι μοναδικός ο ρόλος της και αντικατάστατος. Υπάρχουν χώρες από το Βανκούρβερ μέχρι το Βλαδιβοστόκ, δηλαδή από τη Βόρεια Αμερική, Καναδάς και Ηνωμένε Πολιτείε, τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τη Ρωσία και τα κράτη που προέκυψαν τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Είναι μοναδική λοιπόν για αυτό το λόγο η ΟΑΣΕ και είναι μοναδική επίσης γιατί έχει τρεις διαστάσεις. Πολιτικοστοτιωτική, οικονομική και τη διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως απέδειξε η ιστορία της. Αν κοιτάξουμε τις διάφορες κρίσεις που αντιμετωπίσαμε και η τελευταία στο Κυργιστάν, Πιστεύω ότι η ΟΑΣΕ απέδειξε ότι μπορεί να παίξει ένα ζωτική σημασία ρόλο. Φυσικά ο κόσμος αλλάζει τα τελευταία, τις τελευταίες δεκαετία. Έχουμε μια νέα στρατηγική ε, για την ασφάλεια. Υπάρχουν νέες απειλές, ε, κυβερνοαπειλή, οργανωμένο έγκλημα, εμπορία ανθρώπων, ε, ενεργειακή ασφάλεια και πολλά άλλα θέματα. Και απέναντι σε αυτές τις απειλές μπορεί να παίξει το ρόλο της ΙΟΑΣΕ. Γι' αυτό υπάρχει διαδικασία της Κέρκυρας που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια από, τις, από, τους, από την Ελληνική Προεδρία. Απαντώντας στην πρόσκληση του Ρωσικού Προεδρου Ο πρόεδρος, όπως είπατε, ε, ετοιμάζει αυτή τη σύνοδο κορυφή στην Αστάνα 35 χρόνια μετά την διάσκεψη του Ελσίνκη. Και συμφωνώ πλήρως μαζί σας και θέλω να το συζητήσουμε εδώ ότι θα πρέπει να συζητήσουμε το περιεχόμενο του κειμένου μας. Ποια θα είναι η αντίδρασή μας, η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο της Αστάνας, αλλά και του συγκεκριμένου μας οργάνου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το ψήφισμα λοιπόν τονίζει τη σημασία της διατήρησης της ισορροπίας μεταξύ των τριών διαστάσεων της πολιτικο-στρατιωτικής, της οικονομικής και περιβαλλοντικής και φυσικά της ανθρωπιστικής. Επίσης, όπως είπα, πρέπει να δώσουμε σημασία στην ανάπτυξη περαιτέρω αυτών των διαστάσεων αλλά κυρίως την οικονομική και την περιβαλλοντική. Και για να υπάρξει ενεργειακή ασφάλεια και χάρη στην ΟΑΣΕ, αλλά και για να προωθήσουμε και τα περιβαλλοντικά θέματα. Υπάρχει προστιθέμενη αξία της σταδιωτικής διάστασης. Η ΟΑΣΕ παίζει ένα σημαντικό ρόλο ε, και τον έπαιξε και στο παρελθόν. Η, η σύμβαση για τα όπλα η σύμβαση του 1999. Φυσικά υπάρχουν και κάποια, υπήρξαν και κάποια προβλήματα, κάποια μειο, μειονεκτήματα. Ε, η σύγκρουση στη Γεωργία το 2008 που δεν έχει λυθεί ακόμα, κάποιες παρατεταμένες και ανεπίλητες ε, συγκρούσεις, την ε, υπερνιστερία στον Κάφκασο κτλ. Αλλά αυτή η στρατιωτική διάσταση νομίζω παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι τμήμα και αναφέρεται στο ψηφισμά μας. θα πρέπει να συζητήσουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στην επίτευξη των κοινών αυτών στόχων. Τις σχέσεις μας επίσης και την ε, συνεισφορά του Κοινοβουλίου στην όλη διαδικασία. Επίσης, κατά τη γνώμη μου, και από την προσωπική μου πείρα θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα ενδυναμώσουμε με τη, τη σχέση μας με την κοινοβουλευτική συνέλευση της ΟΑΣΕ. Ίσως θα πρέπει να ενισχύσουμε τη συμμετοχή μας στη συνέλευση αυτή. Και αυτό που προτείνω επίσης στο ψήφισμα είναι το Συμβούλιο ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να έχει μια πρόσκληση στη Σύνοδο και αυτό να το εξασφαλίσει βεβαίως το Συμβούλιο. Εκπροσωπώντας έτσι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη Σύνοδο Παρουσιάζω λοιπόν αυτή τη δήλωση. Είναι ένα ανοιχτό κείμενο. Περιμένω να κάνουμε μια συζήτηση τώρα. Περιμένω τα σχόλιά σας. Έχουμε μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου χρόνο για, τα, για τις τροπολογίες και θα ψηφίσουμε το ψήφισμα αυτό στις 5 Οκτωβρίου. Αυτά. Ευχαριστώ τον κύριο Ρότσεκ. Ο κύριος Σόλτς. Τρία λεπτά. Ähm, Ευχαριστώ για τη δυνατότητα να εκφραστώ σαν σκιώδης εισηγητής επί του θέματος και να παρουσιάσω ορισμένες ανησυχίες. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω για την έκθεση αυτή που βαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, συμβάλλει σε μια συνεργασία όλων των ευρωπαϊκών χωρών σε ένα πνεύμα εμπιστοσύνης ε, που θα είναι προς όφελος όλων. Θα πρέπει να σκεφτούμε εάν το θέμα του ΟΑΣΕ σαν σύστημα ασφαλείας, ε, ένα θέμα δηλαδή το οποίο είχε είχε προκύψει και στο παρελθόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για μελλοντική επίλυση διεθνών ε, διαμαχών και αυτό θα πρέπει να ε, προωθηθεί και κατά την ε, Προεδρία του Καζάρα διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει διάφορες διαμάχες ε, στην Ευρωπαϊκή Ήπερο Ήπειρο ε, όπου ένας ε, ειρηνικός μηχανισμός θα είναι χρήσιμος και ε, αναφέρθηκαν και στην έκθεση οι διάφορες διαμάχες του παρελθόντος. Όσον αφορά το περιβάλλον θα πρέπει να σκεφτούμε και πάλι εάν δεν μπορεί ο μηχανισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιηθεί από κοινού ή στο μέλλον για την προστασία του περιβάλλοντος ε, και ε, για την αντιμετώπιση των κλιματολογικών αλλαγών. Έχω όμως διαφορετική αντιμετώπιση όσον αφορά τις σχέσεις ε, των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ. Σε, κατά τη συζήτηση πρέπει να σκεφτούμε αν όντως μπορεί ο ΑΣΕ να χρησιμοποιήσει χρησιμοποιηθεί ε, δεσμευτικά για να εκπροσωπήσει ευρωπαϊκές χώρες και να αποδυναμώσει το ΝΑΤΟ. Ευχαριστώ. Κυρίλοφ, τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ θερμά τον Λίμπο για την έκθεσή του πολύ ισορροπημένη και επίκαιρη γιατί μας δίνει πολλές ιδέες για την ανάγκη του ρόλου της ΟΑΣΕ. Γιατί με τις εξελίξεις των τελευταίων ετών αποδυναμώθηκε κάπως ο ρόλος της. Θα πρέπει λοιπόν να συμμετέχουμε ενεργά στην ενίσχυση του ρόλου του ΟΑΣΕ, ιδιαίτερα μετά τη θέση ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας, ώστε να ενδυναμωθεί η οργάνωση αυτή. Αυτά γενικά. Τώρα έρχομαι στα πιο συγκεκριμένα. Για την ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ απτά και πιστικά ο κύριος Ρόουτσεκ μας μίλησε για την για τον ισχυρό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν θα πρέπει να αποδυναμώσει το ρόλο της ΟΑΣΕ, αντίθετα θα πρέπει να τον ενισχύσει. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ισχύει και για τα κράτη-μέλη της ΟΑΣΕ. Η πολιτικοστρατιωτική διάσταση είναι αρκετά σημαντική και σε μερικούς τομείς δημιουργεί προβληματισμό. Σωστά αναφέρεται στην παράγραφο 6 ότι υπάρχουν εκκρεμείς διενέξεις και διδαχθήκαμε από το πάθημα του 2008 από την ρωσικο-γεωργιανή σύγκρουση, αλλά και με το, την παγωμένη σύγκρουση του Ναγκόρνο Καραμπάχ και της υπερθετινιστερίας. Είναι προβληματική κατάσταση στον Κάφκασο και γι' αυτό χρειαζόμαστε και ισχυρό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και ενίσχυση του ρόλου της ΟΑΣΕ και καλό θα ήταν να ληφθούν και πρωτοβουλίες στην περιοχή του Καφκάσου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά την ε, οικονομική διάσταση της ΟΑΣΕ θα πρέπει να μιλήσουμε και για την παράγραφο 10 και να ενισχύσουμε την διαπεριφερειακή συνεργασία μεταξύ των χωρών. Έτσι θα εμπεδοθεί και η εμπιστοσύνη μεταξύ τους. Γιατί πολλές φορές οι χώρες αυτές είτε για ιστορικούς λόγους είτε για τις εξαιτία των εκκρεμών, συγκρούσεων δεν έχουν το κουράγιο να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη μεταξύ τους. Νομίζω ότι καλό θα είναι να δημιουργηθεί ένα πρόσφορο και αίσιο κλίμα για την αποκλιμάκωση των εντάσεων και για την εδραίωση της ε, εμπιστοσύνης μεταξύ τους. Πολύ σωστά αναφέρει ο εισηγητής και το θέμα τους, των εκτοπιστέντων και των προσφύγων. Είναι εκατομμύρια αυτοί οι άνθρωποι. Οι εσωτερικά εκτοπιστέντες και οι πρόσφυγες. Θα πρέπει λοιπόν να συμβάλλουμε στην ενίσχυση του ρόλου της ΟΑΣΕ, αλλά το πιο σημαντικό είναι, δεδομένων των νέων αρμοδιοτήτων που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, να αναλάβουμε περισσότερες ευθύνες και να συμμετέχουμε πιο δραστήρια. Η ομάδα του Μίνσκ είναι κάτι σημαντικό, ήδη το υπογραμμίσαμε, θα πρέπει να υπάρξει εντολή συγκεκριμένη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε κύριε Κυριλόφ. Για τρία λεπτά το λόγο έχει ο κύριος Γκζίμπ. Ευχαριστώ. Τα τελευταία δύο χρόνια είχαμε πολύ εντυπωσιακές εξελίξεις και σημαντικά γεγονότα που υπογραμμίστηκαν και στην έκθεση ε, από τον εισηγητή τον κύριο Ρότσακ και είναι πολύ ε, σημαντικές αυτές οι εξελίξεις. Για παράδειγμα, η έναρξη της διακασίας αυτής ε, της Κέρκυρας με πρωτοβουλία του προ... Ρώσου Προέδρου Ματιου Βιέντεφ. Είχαμε και την συνδιάσκεψη της ε, Βιέννης και τον Ιούλιο πρόσφατα την Υπουργική Διάσκεψη της ε, ΟΑΣΕ που ουσιαστικά δίνουν συνέχεια στην αρχική πρωτοβουλία της Κέρκυρας. Η πρωτοβουλία της Κέρκυρας ε, φύσηξε νέο αέρα στην κατάσταση αυτή και αυτή η νέα πνοή θα πρέπει να αξιοποιηθεί και να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα αυτής της σημαντικής οργάνωσης ασφάλειας και συνεργασίας στην Ευρώπη. Αλλά θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να αντιδράσουμε και απέναντι στις νέες απειλές που επισημαίνονται σωστά στο, στο σχέδιο του ψηφίσματος. Για το θέμα της κοινή ασφάλειας είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει όμως ε, και το σημαντικό θέμα της συνθήκης ε, των σημαντικών όπλων. Η διαδικασία της Κέρκυρας πλαισιώνεται κυρίως από την ΟΑΣΕ αλλά άπτεται πολύ σημαντικών πτυχών της ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει και κάποιες νέες προτάσεις. Η γενική πάντως συζήτηση είναι θετική. Θα πρέπει πολύ ρεαλιστικά να προσεγγίσουμε και να επιδιώξουμε την επίλυση σημαντικών προβλημάτων. Ο διάλογος θα πρέπει να συνεχιστεί και να είναι πολυδιάστατος. Να μην επικεντρωθεί όπως επιχειρούν ορισμένες χώρες να επικεντρωθεί η προσοχή της συζήτησης στο θέμα της ε, hard security, όπως λέμε, αλλά να περιλάβει η συζήτηση και τα θέματα του soft security, όχι μόνο της ε, σκληρής ασφάλειας, αλλά και της ήπιας ασφάλειας. Επίσης, η τι συνέβη με την Προεδρία του Καζακστάν. Νομίζω ότι ήταν αρκετά επιτυχημένη η Προεδρία του Καζακστάν και καλό θα ήταν να διαμορφωθεί μία ισχυρή σε διάταξη. Θα ήταν κρίμα μετά τη διάσκεψη κορυφής να μην υπάρξουν απτά αποτελέσματα και να μην ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις. Επίσης θα πρέπει να διαμορφωθεί μια εντολή με τη μορφή σχεδίου δράσης για την οργάνωση αυτή. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών για τα θέματα αυτά. Σε ό,τι αφορά την υπουργική διάσκεψη του Υπουργικού Συμβουλίου δηλαδή, αλλά και άλλες ε, συνεδριάσεις που έγιναν, υπάρχει αισθητή η άξη της ε, σημασίας της ΟΑΣΕ. Και αυτό το θέμα, δηλαδή της ενίσχυσης της σπουδαιότητας της ΟΑΣΕ, θα πρέπει να υπογραμμιστεί στο ψήφισμά μας. Και το τελευταίο μου σχόλιο. Έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να προωθήσουμε αυτή τη διαδικασία ώστε η διάσκεψη κορυφής να φέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Γιατί αν δεν ε, καταλήξουμε σε αυτά αποτελέσματα, ίσως διακυβευτεί το ίδιο το μέλλον της ΟΑΣΕ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Γκζιμπ. Το λόγο κύριο Στάνοφ για τρία λεπτά. Ευχαριστώ uh, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ισοσκελισμένη έκθεση. Πριν από μερικά χρόνια είχα στηρίξει την κίνηση να ε, ε, προτείνουμε την Καζακική Προεδρία στον ΟΑΣΕ και χαίρομαι που επέτυχαν το στόχο τους. Είναι ενδιαφέρον θεσμός ο ΟΑΣΕ. Δεν θέλω να υπερβάλλω τη σημασία αλλά υπάρχει διαμάχη μεταξύ του ρόλου ασφαλείας και της προφανούς προσπαθίας να προβάλλουν την δημοκρατία. Ε, είμαι υπέρ της δημοκρατίας και ιδίως κατά την ε, πορτοκαλί ε, επανάσταση στην ε, Ουγγαρία είχα παρατηρήσει ε, ε, πόσο είχαν στηριχθεί οι διεφθαρμένες εκλογές τις οποίες είχαμε ε, παρακολουθήσει σαν βουλευτές εκείνη την εποχή. Ε, δεν ε, είναι πολύ δημοκρατικά τα κράτη της κεντρικής Ευρώπης αλλά υπάρχει μία μοναδική δομή πολυμερής και βλέπουμε στην κεντρική Ασία μία αναδιόμενη περιοχή διαμαχών για, ε, που, από χώρες που επιζητούν την, να υπερισχύσουν τον άλλον και ε, εξουδετερώνουν μεταξύ τους την ε, εχθρικές κινήσεις εναντίον των δυτικών συμφερόντων στην Κεντρική Ασία η χώρα ε, της Προεδρίας δεν είναι πολύ δημοκρατική αλλά είχε στηρίξει τη διαμάχη στη Μολδαβία και στην ε, Τρανσνιστρία. Ε, ήθελα να σας πω ότι όταν έχουμε εκλογικές παρα... εκλογικούς παρατηρητές οι οποίοι αποστέλλονται από το Κοινοβούλιο υπάρχει μία τριμερής διαμόρφωση ε, από το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον ΟΑΣΕ και την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλαδή, το οποίο όμω πάντοτε είναι σε μειονεκτική θέση διότι το ΟΑΣΕ αυτομάτως ε, προεδρεύει και παρουσιάζει την τελική έκθεση στη σελίδα σελίδα 24 αναφέρονται οι σχέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τον ΟΑΣΕ πράγμα το οποίο δεν παρουσιάζει γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντοτε πρέπει να είναι σε μειονεκτική θέση στις αποστολές όταν πηγαίνουμε ε, σαν παρατηρητές στις χώρες του ΟΑΣΕ. Ευχαριστώ. Τον ρόλο για τα τελευταία σχόλια έχει ο κύριος Ράουτσεκ. ο εισηγητής δηλαδή. Ευχαριστώ. Ε, σημείο προς σημείο ε, θα ήθελα να επανέλθω στα διάφορα θέματα. Ο κύριος ε, Σούλτς και ο κύριος Τάνοκ ανέφεραν την κεντρική, την κεντρική Ασία είναι μια περιοχή όπου ο ΑΣΕ μπορεί και θα έπρεπε να παίζει μεγαλύτερο ρόλο και αυτό απεδείχθηκε με την Καζακική Προεδρία. Γιατί δηλαδή το Καζακστάν αυτή τη στιγμή ανέλαβε την Προεδρία. Υπάρχουν προσμονές οι οποίες ήταν πολύ υψηλές και ο ρόλος αυτός ανατέθηκε ή στο Καζακστάν για να μπορέσει να αναβαθμίσει τη θέση του. Είναι σημαντικό λοιπόν και γι' αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε στην έκθεσή μας και στη σύστασή μας. διότι δεν αναφερόμαστε μόνο στην Κεντρική Ασία αλλά ε, υπάρχουν και ορισμένα θέματα τα οποία εμπλέκονται το Αφγανιστάν, το Πακιστάν αν κοιτάξουμε δηλαδή το χάρτη της περιοχής είναι μια περιοχή πολύ σημαντική ο κύριος Σόλτς επίσης αναφέρθηκε στην προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος και πιστεύω ότι η διάσταση αυτή στο μέλλον θα έχει όλο και μεγαλύτερη σημασία. Εάν λοιπόν έχετε κάποια πρόταση όσον αφορά κάποια τροπολογία, σας ακούω. Όταν είπατε ε, ε, εκεί όμως που εγώ διαφωνώ μαζί σας είναι ο ρόλος του ΝΑΤΟ. Ναι μεν τονίζεται ότι είναι προς ε, όφελόν μας να ενισχύσουμε τον ΟΑΣΕ και να ενισχύσουμε τη θέση Ευρωπαϊκής Ενώσεως ιδίως μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας και ε, τα νέα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Δεν πιστεύω όμως ότι μας ωφελεί να αποδυναμώσουμε τον ρόλο άλλων θεσμικών οργάνων και ιδιαιτέρως του ΝΑΤΟ. Διότι το ΝΑΤΟ ακόμη ε, διαδραματίζει ένα πολύ σοβαρό ρόλο όσον αφορά την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και κανείς άλλος δεν μπορεί να αναλάβει το ρόλο αυτό. Βεβαίως, το ΝΑΤΟ δεν είναι ένας οργανισμός εξοπλισμένος για να επέμβει στην Κεντρική Ασία αλλά εάν ο ΑΣΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ορισμένες δυνάμεις του ΝΑΤΟ θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους τους οποίους επιζητεί ο ΑΣΕ και προσπαθεί να επιτύχει. Ο κύριος Κυρίλοφ αναφέρθηκε στην περιφερειακή συνεργασία. Δεν είμαι αντίθετος στην περιφερειακή συνεργασία διότι η οικονομική περιφερειακή συνεργασία μπορεί όχι μόνο να ε, συμβάλλει στον οικονομικό ρόλο αλλά μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση των ε, σχέσεων μεταξύ των λαών στην ανάπτυξη του τουρισμού αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι σε μια τόσο μεγάλη περιοχή από το Βανκούβερ στο Βλαδιβοστόκ είναι πάρα πολύ δύσκολο να οριοθετήσουμε την περιοχή αυτή θα έπρεπε όμως αναφερθεί ε, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της οργανώσεως συμφωνώ πολλές φορές ε, ενοχλούμεθα και άλλα μέλη του ΑΣΕΑ ενοχλούνται διότι ορισμένες ε, εργασίες όσον αφορά την ανάλυση των ε, διαμαχών στον Αγκόρνο Παραγκά, ε, στην Τρανσνιστρία και ούτω καθεξής δεν παρουσιάζονται σωστά και θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας προς αυτή την κατεύθυνση. Είπατε επίσης ότι δεν ασχολόμαστε μόνο με την ε, ασφάλεια, με τη σκληρή έννοια αλλά και με την, τους νέους τους κινδύνους για την ασφάλεια και πιστεύουμε ότι η ανθρώπινη διάσταση είναι πολύ σημαντική. Και γι' αυτό για να απαντήσω και στον κύριο Τάνοκ θα ήθελα να πω ότι εάν αναπτύξουμε τη δημοκρατία, τα πολιτικά δικαιώματα των πολιτών, ε, εκτελούμε μία διεργασία που συμβάλλει ε, την ε, ενίσχυση του και ενισχύουν αυτή τη διαδικασία διότι πολλοί δεν επρόκειτο να είναι εδώ εάν ε, δεν ε, είχε υπάρξει η πράξη του ο Ελσίνκι του 75 και προσβλέπω εις τους ο, Πολωνούς και Τσέχους συναδέλφους οι οποίοι συνέβαλαν στην πτώση του κομμουνισμού και στην ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ιδέας της δημοκρατίας. Είναι δηλαδή κάτι πολύ σημαντικό και ένας πολύ βασικός ρόλος για τον ΟΑΣΕ διότι όλα τα κράτη-μέλη του ΟΑΣΕ δεν είναι απολύτως δημοκρατικά ε, μπορέσαμε να επιτύχουμε ορισμένα αποτελέσματα και ουσιαστικά αυτό χρειάζεται ο ΟΑΣΕ και αυτή θα πρέπει να είναι και η προσπάθειά μας. Συλλογικά λοιπόν ας κοιτάξουμε στις επόμενες εβδομάδες τι συγκεκριμένα προγράμματα έχουμε, τι συγκεκριμένες προτάσεις μπορούμε να διατυπώσουμε κατά τρόπον ώστε κατά τη διάσκεψη κορυφής και πριν αυτή να μπορέσουμε να συμβάλλουμε εις ε, την συζήτηση, να την κάνουμε πιο συγκεκριμένη. Ε, ε επίσης ε, ο, ο ΑΣΕ είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός Κανείς δεν μπορεί ή δεν θα έπρεπε να επηρεάζει την ανεξαρτησία του γιατί έχει ένα βασικό ρόλο για την πρόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τον εκδημοκρατισμό, τον ρόλο των μειονοτήτων διότι αν κοιτάξουμε την μετασοβιετική κατάσταση στο χώρο της Κεντρικής Ασίας ή το θέμα των πληθυσμών των τον ε, Ρώμα στο χώρο μας ε, επίσης επηρεάζει. Όσον αφορά τις, ε, τις αποστολές παρατηρητών ή τις εκλογές γιατί έχουμε το μειονεκτικό ρόλο. Είναι επίσης μέρος της ιδέας μας. Πρέπει να ενισχύσουμε το ρόλο μας στον ΟΑΣΕ. Γι' αυτό και θα έπρεπε να αναλάβουμε μεγαλύτερο ρόλο στην κοινοβουλευτική συνέλευση και κατά αυτόν τον τρόπο σιγά σιγά θα μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε το ρόλο μας όσον αφορά τη διαδικασία παρακολούθησης των εκλογών. Σας ευχαριστώ όμως όλους για τη συνδρομή σας. Ε, προσβλέπω στις τροπολογίες σας και όπως σας είπα η ε, προθεσμία λήγει στις 14 ε, Σεπτεμβρίου το μεσημέρι. Εκτός προγράμματος ο κύριος Σόλτς θέλει να παρέμβει για δύο λεφτά. Κύριε Πρόεδρε, είχα ζητήσει το λόγο και προηγουμένως, αλλά ίσως ε, δεν με είδατε. Αν λοιπόν υπάρχει χρόνο θα ήθελα να πω ότι θεωρώ ότι το σχέδιο αυτό ψηφίσματος είναι πολύ σημαντικό, διότι ε, ο ρόλος εργασίας του ΟΑΣΕ στις τρεις διαστάσεις του επιβεβαιώνεται και καταγράφεται. Ε, το σχέδιο αυτό ψηφίσματος ε, στηρίζει ε, και την προσπάθεια με Μετβεντέφ να στηρίξει τη διαδικασία της Κερκύρας αλλά όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μας οι οποίοι ε, θέλουμε να βελτιωθεί και να βασιστεί η εργασία του ΟΑΣΕ έχω την εντύπωση ότι οι Ρώσοι προσπαθούν να καπελώσουν τον ΟΑΣΕ και αυτό θα έπρεπε να το κατακρίνουμε διότι θεωρώ ότι ο ρόλος της Ρωσίας όσο και να είναι βασικό να είναι ε, η Ρωσία και οι πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες στον ΟΑΣΕ και να ε, συζητούν ε, αυτές τις διαμάχες δεν είναι θετικός ο ρόλος αυτός της Ρωσίας στον ΟΑΣΕ. Το είδαμε στην Τσετσενία και στις τελευταίες τελευταίες δημοτικές εκλογές οι οποίες ήταν διεφθαρμένες και αυτό παραδέχτηκε και ο Ρώσος πρόεδρος. Ε, θα έπρεπε λοιπόν να αξιολογούμε κριτικά το γεγονός ότι ε, οι Ρώσοι ζητούν να συμβάλλουν ε, περισσότερο στα πλαίσια του ΟΑΣΕ. Ίσως είναι κάτι λοιπόν το οποίο μπορεί να περιληφθεί σε μία τροπολογία και ελπίζω ότι θα με στηρίξετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σούλτς. Ο εισηγητής θέλει να προσθέσει κάτι, να απαντήσει. Συμφωνώ πλήρως, συμφωνώ πλήρως. Αυτή είναι η απάντησή μας. Σύντομη και αποτελεσματική απάντηση. Τώρα, για το χρονοδιάγραμμα αυτής της έκθεσης, όπως ε, Σα είπαν στις 14 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι είναι τελική προθεσμία για την παρουσίαση των τροπολογιών και 5 Οκτωβρίου θα γίνει η συζήτηση των τροπολογιών και η ψήφισή τους στην Επιτροπή. Η ψήφιση στην ε, Ολομέλεια θα γίνει στη δεύτερη Ολομέλεια του Οκτωβρίου, λέει ο Πρόεδρος. Πάμε Τώρα, στο επόμενο σημείο που αφορά τη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο προπολογισμού για το 2011, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο. Όλα τα τμήματά του. Ο πρωταγωνιστής αυτής της έκθεσης είναι ο κύριος Αλαφράνκα. Είναι ο εισηγητής. Έχουν κατατεθεί 87 τροπολογίες. Και μετά την παρουσίαση του κυρίου Σαλαφράνκα, θα ακούσουμε τους σκιώδεις εισηγητές και τους συντάκτες των τροπολογιών για να μας εξηγήσουν γιατί ακριβώς ζητούν αυτές τις τροπολογίες. Κύριε Σαλαφράγκα, παρουσιάστε μας το κείμενο. Eh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα εν συντομία, πριν περάσουμε στο κυρίως θέμα, να υπενθυμίσω το δημοσιονομικό πλαίσιο και ιστορικό της ε, κατηγορίας 4 που μας ενδιαφέρει άμεσα. Προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αύξηση 5,56% σε ό,τι αφορά της ε, αναλήψεις υποχρεώσεων, κάτι που προϋποθέτει για την ε, διακυριστική χρήση του 2011 2 800 εκατομμυρίων. Σε ό,τι αφορά την τέταρτη κατηγορία, ο γενικός προϋπολογισμός του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκε μόνο κατά 0,76%, 77%. Κάτι που δείχνει σαφέστατα τις ε, ελλείψεις και τις αδυναμίες που αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο όταν προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε σε εξωτερικές μας υποχρεώσεις που είτε είναι προβλέψιμες είτε προσδόκητες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σχέδιο του προϋπολογισμού προτείνει σημαντική αύξηση για την ε, ανταπόκριση της κρίσης, για το σύμφωνο σταθερότητας 25% ε, επιπλέον, ε, στην ΚΕΠΑ συν 16%, πολιτική γειτονία συν 19%, ε, για, το ε, για την Ανατολή και για το Νότο 6,6% και στην ανασυγκρότηση του Αφγανιστάν με βάση τις ε, δεσμεύσεις που λάβαμε στη, στη των δωρητών συν 25%. Επίσης προβλέπονται σημαντικές μειώσεις. Για παράδειγμα, στην πολιτική ενίσχυση προς την Παλαιστίνη περιστολή κατά 95 εκατομμύρια σε ό,τι αφορά τις αποστολές παρατήρησης εκλογών. Αναφέρθηκε στην προηγούμενη συζήτηση. Και μάλιστα μετά τις διαπραγματεύσεις που είχε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τα λοιπά θεσμικά όργανα. Όχι μόνο έχουμε την Προεδρία στις ε, ε, αποστολές παρατήρησης, αλλά και ε, μεγάλη πρωτοβουλία και ταυτόχρονα θα συμμετέχουμε στο διορισμό των επικεφαλή επικεφαλής αυτών των αποστολών. Αλλά και σε άλλα κεφάλαια έχουμε σημαντικές μειώσεις σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με κάποιες χώρες. Ιράκ, Ιράν, Ιεμένη, συνολική μείωση 16% για τη συνεργασία με τις χώρες αυτές. Μετά την παρουσίαση αυτού του σχεδίου προϋπολογισμού τη Επιτροπή, το, Ευρωπαϊκό, το Συμβούλιο ε, πρότεινε μια πολύ αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία και δραστικές ε, μειώσεις σε όλε τι επιχειρησιακέ γραμμέ σε κατά 100 εκατομμύρια ευρώ και επίση στι διάφορε κατηγορίε ε, που αφορούν την διοικητική υποστήριξη των επιχειρησιακών ε, δημοσιονομικών γραμμών επίσης πρότεινε μείωση. Επίσης προτάθηκε αύξηση του αποθεματικού κατά 70 μόνο εκατομμύρια, για το, από το 70 εκατομμύρια σε 164 εκατομμύρια για το 2011 και ταυτόχρονα το Συμβούλιο πρότεινε μια πολιτική ελέγχου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μειώνοντας δραστικά τις πιστώσεις πληρωμών κατά, σε ύψος 591 εκατομμυρίων. Αυτή ήταν η μείωση που πρότεινε το Συμβούλιο για τις πιστώσει πληρωμών. Με το σχέδιο ψηφίσματο που έχετε λάβει στου φακέλου σα, εγώ επισημαίνω την ανάγκη εξασφάλιση των εξωτερικών δράσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, φυσικά τηρώντα τι ανηλυμένε υποχρεώσει μα και δεσμεύσει. Επίση, η σύσταση τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική δράση θα πρέπει να ε, συνοδευτεί με τα κατάλληλα επιχειρησιακά κονδύλια. Και όλα αυτά θα πρέπει φυσικά να τα συνδυάσουμε με τα στοιχεία και τις απαιτήσει της δημοσιονομικής πειθαρχία. Η δημοσιονομική διαδικασία είναι μια διαδικασία που ολοκληρώνεται στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Θα μπορούσα εγώ να ακολουθήσω μια πολιτική ανοίγματο τεράστιου και διαλλακτικότητα και να πω ότι δέχομαι όλες τις τροπολογίες των συναδέλφων, αλλά αυτό είναι πανεύκολο για να το πει κανείς, αλλά δεν είναι και πολύ υπεύθυνο ή σοβαρό. Θέλουμε να λάβουμε υπόψη τις πιο σημαντικές ανησυχίες και προβληματισμούς, αλλά ε, έχοντας υπόψη την ανάγκη δημοσιονομική πειθαρχία. Επίσης, αν ξεφύγουμε, αν παρεκκλίνουμε από τις δημοσιονομικές ισορροπίες και προβλέψουμε σημαντική αύξηση βάση τροπολογία, ούτω ή άλλω τελικό λόγο θα τον έχει η Επιτροπή Προπολογισμών και αυτή θα προβεί σε δραστικέ μειώσει, αδιαφορώντα για τι δικέ μα προτεραιότητε. Γι' αυτό λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, και επειδή δεν θέλω να μακρηγορήσω, προτιμώ να ακούσω τι ε, ανησυχίε των συναδέλφων, θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Σε ό,τι αφορά το σχέδιο ψηφίσματο, υπευλήθησαν 7 τροπολογίε. Μπορώ να δεχτώ τι περισσότερε από αυτέ γιατί είναι λογικέ. Ε, η κυρία Μπραντ που είναι παρούσα υπέβαλε τη δεύτερη τροπολογία θέλει να δώσει έμφαση στην πρόληψη των συγκρούσεων. Συμφωνώ με την τροπολογία 2 αρκεί να μην ξεφύγουμε από τα όρια και τα πλαίσια μας. Η πολιτική εξωτερικών δράσεων της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης θα πρέπει φυσικά να λάβει υπόψη και την ανάγκη πρόληψης των συγκρούσεων, αλλά δεν είναι αυτή η ύψιστη προτεραιότητα. Πάντως θα το λάβω υπόψη με μια προφορική τροπολογία μου για να εισακουστεί η ανησυχία σας ε, για την ανάγκη λήψη υπόψη της πρόληψης των συγκρούσεων. Κύριε Γουαλτιέρη, και εσείς καταθέσατε δύο τροπολογίες. Η μία αφορά την ανάγκη δημοσιονομικής πειθαρχία και λιτότητας. Καταρχήν να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Γουαλτιέρη για την συνεργασία του, γιατί συνυπογράψαμε μία σειρά τροπολογιών, οπότε και εγώ μπορώ να δεχτώ τις δικές του τροπολογίες, αρκεί φυσικά να μην ξεπεράσουμε τα όρια της συμβαστικής μας ε, συμφωνίας και την τροπολογία κούκανου θα μπορούσα να δεχτώ. Και ε, ερχόμαστε στο κυρίω θέμα, τι τροπολογίε που επιβεβαιώνουν τα ποσά. Γιατί όταν μιλούμε για προπολογισμό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα ποσά, τα συγκεκριμένα κονδύλια. Κατατέθηκαν 52 τροπολογίε πέραν των 34 που συνυπογράψαμε με τον κύριο Γουαλτιέρη και από αυτέ τι 52 τροπολογίε που κατατέθηκαν ένα μεγάλο τμήμα τους και οι περισσότερες ανησυχίες τους, το 80% θα έλεγα των ανησυχιών, καλύπτονται από τις κοινέ μας τροπολογίες με τον κύριο Γουαλτιέρη. Για τα πιο σημαντικά θέματα, και αν θέλετε μετά μιλούμε για τις λεπτομέρειες, είναι η σημαντική προτεραιότητα που δίνουμε, όπως συζητά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την χρηματοδότηση, επαρκή χρηματοδότηση της ε, ΚΕΠΑ, αλλά σε ό,τι αφορά τα έκτακτα μέτρα, που πραγματικά είναι το πιο αφιλεγόμενο σημείο, για να διαφυλάξουμε τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους όρους της συμφωνίας στην οποία κατέληξαν η Μπροκ, Γουαλτιέρη και Φερχόφστατ σε ό,τι αφορά την υπηρεσία εξωτερικών δράσεων, θα πρέπει πρώτα να καθοριστούν τα μέτρα διαφάνειας για τη σχέση μεταξύ των θεσμικών οργάνων σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του προπολογισμού. Προ το παρόν, προτείνω να αφήσουμε αυτό το κονδύλιο στο αποθεματικό, μέχρι ότου εξασφαλιστεί δυνατότητα διενέργεια επαρκού ελέγχου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προτείναμε σημαντική αύξηση των ε, ποσών για τι δράσει υποστήριξη τη Παλαιστινιακή Αρχή. Νομίζω ότι είναι σκόπιμο κάτι τέτοιο, γιατί τώρα αρχίζουν οι διαπραγματεύσει, οι ειρηνευτικέ διαπραγματεύσει στη Μέση Ανατολή. Και μάλιστα από διαβουλεύσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι προβλέψεις της ε, υστερούν σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες, γι' αυτό και πρότεινα αύξηση των σχετικών κονδύλιων. Σε ό,τι αφορά τις αποστολές παρατήρησης εκλογών, όπως είπα και προηγουμένως, αυτό το μέσο είναι από τα πιο σημαντικά που διαθέτει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι επικεφαλής των αποστολών είναι ευρωβουλευτές και μάλιστα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει και στο διορισμό των εκπροσώπων Οπότε νομίζω ότι δεν είναι προς το συμφέρον μας ε, ε, και ιδιαίτερα των αποστολών να μειώσουμε τα κονδύλια σε σχέση με προηγούμενες ε, διαχειριστικές χρήσεις. Δεν θα ήθελα να υπερβώ το όριο των 5% αλλά να τονίσω τη σημασία που έχουν τέτοιες δράσεις παρατήρησης εκλογών για το Κοινοβούλιο. Σε ό,τι αφορά την γραμμή για το μέσο προάσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο, ούτε και αυτή η γραμμή θα πρέπει να μειωθεί, ούτε ως προς τις διοικητικές δαπάνες, ούτε ως προς τα σχόλια για τις δημοσιονομικές γραμμές. Και εκεί επαναφέραμε το σύνολο του ποσού. Υπάρχει και το θέμα των διοικητικών δαπανών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μείωση 24 εκατομμύρια. Τελικά περιοριστήκαμε σε 7,5 εκατομμύρια μείωση. Είναι λογική αυτή η μείωση των 7,5 εκατομμυρίων γιατί κατά 70% επανήλθαμε στην αρχική πρόταση προσπαθώντας να διαφυλάξουμε και την αξιοπιστία μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε όλα τα πιλωτικά προγράμματα που υπέβαλαν τότε οι σκιώδεις ηγητές και από την άποψη αυτή η κυρία Γιάτερ Μάκη κατέθεσε και κάποιες ε, τροπολογίες για σχέδια. Θα ήθελα να επισημάνω ότι αυτή τη στιγμή είναι δυσάρεστο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει υποβάλει τον προϋπολογισμό της για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Γιατί όλη αυτή η προσπάθεια που κάνουμε για τη διαχειριστική χρήση του 2011 θα εξαρτηθεί από τη λύση που θα δοθεί για την ΕΑΣ θα πρέπει να αποφύγουμε επικαλύψεις. Γιατί αν δεν διαθετηθεί πρώτα το θέμα της εξωτερικής υπηρεσίας, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, θα είναι αναπόφευκτες οι επικαλύψεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά διάφορες άλλες τροπολογίες. Καταρχήν, η τροπολογία 50.03 της κυρίας Χάουταλα, που ζητά την πρόβλεψη ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Θιβέτ. Εγώ έχω προσωπική γνώμη, αλλά θέλω και τη δική σας αντίδραση. Υπάρχει μια πολύ σημαντική τροπολογία της κυρίας Φλότρ και εκεί έχω διαμορφωμένη γνώμη, αλλά περιμένω και τη δική σας αντίδραση και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η κυρία Φλότρ προτείνει να μπουν 6 εκατομμύρια στο αποθεματικό για τη δικαστική συνεργασία με την Ισία, προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στην Ισία. Και τέλος η κυρία Μπραντνερ προτείνει την τροπολογία 5037 που κάνει λόγο για προπαρασκευαστική δράση εν ώψη της σύστασης μιας ομάδας διαμεσολάβησης για την σύσταση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Ξέρω ότι η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού κατάρτισε έκθεση για την δημοσιονομική διαχείριση που δεν ε, εξασφαλίζεται από την ΕΑΣ. Ποια είναι τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το σημείο αυτό. Αυτά κύριε Πρόεδρε και περιμένω τα σχόλια των συναδέλφων και μέχρι την ε, ψηφοφορία της Δευτέρας θα προσπαθήσω να λάβω υπόψη όσο δυνατόν περισσότερες ε, τροπολογίες κατατεθούν αρκεί φυσικά να μην διαταραχθεί όπως είπα η ανάγκη αυστηρότητας και λιτότητας αλλά ταυτόχρονα και διαλλακτικότητας προκειμένου να εισακουστούν οι ανησυχίε των συναδέλφων. Πάντω και ω προ το πνεύμα και ω προ το γράμμα του, περισσότερε ανησυχίε νομίζω έχουν καλυφθεί από τι κοινέ μα τροπολογίε με τον κύριο Γουαλτιέρη. Ευχαριστώ κύριε Σαλαφράγκα. Ξεκινάει η συζήτηση. Τώρα θα δώσω το λόγο καταρχά στου σκιώδει εισηγητέ. Και εν συνεχεία θα δώσω στου υπόλοιπου ομιλητέ. Ο κ. Γκουαλτιέρη για τρία λεπτά. Είναι σκιώδη εισηγητή των σοσιαλιστών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σαλαφράγκα για τη δουλειά σας, για την προσπάθειά σας, για την διάθεσή σας να υπάρξει διάλογος, να συνεργαστούμε, που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό σε μια τόσο κρίσιμη πολιτική και οικονομική συγκυρία για τη δράση εξωτερική, την εξωτερική δράση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλό είναι λοιπόν να δοθεί ένα σαφές μήνυμα. Τα νούμερα μας τα παρουσίασε ο κύριος Σαλαφράνκα, δεν θα επανέλθω. Είχαμε εκφράσει κάποιες ανησυχίες για τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδίως για το σημείο που φούρσε την Παλαιστίνη και για το πολύ μικρό περιθώριο που προβλέπεται. Και προφανώς η παρέμβαση του Συμβουλίου ε, μείωσε δραματικά αυτά τα ποσά, χειροτέρευσε την κατάσταση. Και μάλιστα είναι ιδιάζουσα αυτή η ιστορία, γιατί αυξάνονται οι πληρωμές συνολικά του προϋπολογισμού. Αλλά αν δεχτούμε αυτά που λέει το Συμβούλιο, τότε έχουμε μια συνολική περικοπή των πληρωμών του τίτλου 4 κατά 10%. Τι νόημα έχει αυτό. Αυτό που λέει το κείμενο του Συμβουλίου δεν είναι σωστό ότι υπάρχει μια αναλογική περικοπή σε, όλες, σε όλους τους τίτλους. Όχι. Ε, οι περικοπές αυτές ε, αφορούν συγκεκριμένους τίτλους, ε, είναι δυσανάλογες και επομένως ο προπολογισμό δεν είναι σοβαρός και δεν είναι αξιόπιστος με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, με τέτοιες παρεμβάσεις και, του Συμβουλίου και με παρεμβάσεις στο σύμφωνο, στο μέσο μάλλον το προενταξιακό, δεν νομίζω ότι εξασφαλίζουμε την αξιοπιστία της Ένωσης. Πρέπει όμως να είμαστε αξιόπιστοι στη χρήση των πόρων μας και στην χρήση αυτών των χρηματοδοτικών μέσων. Η παρέμβαση συνολικά του Συμβουλίου πιστεύω ήταν αρνητική. Φυσικά, λαμβάνω υπόψη μου τη δύσκολη συγκυρία, το δύσκολο πλαίσιο με στο οποίο λειτουργούμε. Έγινε μια προσπάθεια λοιπόν μέσα σε αυτό το πλαίσιο να επανέλθουμε σε ένα αποδεκτό επίπεδο δεσμεύσεων για τις βασικές προτεραιότητες της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το πνεύμα των τροπολογιών που αφορούν όλες τις περικοπές οποίες προέβη το Συμβούλιο. Και προσπαθούμε να διασώσουμε και να επανέλθουμε στον προϋπολογισμό που είχε προτείνει η Κομισιόν, ιδίως ε, το σημείο που αφορά την Παλαιστίνη. Έχουμε τη Συμφωνία της Μαδρίτης για το, τη δομή του προϋπολογισμού της Αλίας. Ε, είναι σημαντικό ήδη ε, στον προϋπολογισμό του 2011 να υπάρχουν οι γραμμές για τις βασικές, τα βασικά σημεία του προϋπολογισμού της Αλίας. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό που είπε ο κ. Ε, Σαλαφράγκα για τι τις για το Θιβέτ και αυτό που είπε για την, ε, την Ισία και αυτό συζητήσιμο είναι, για να το πω έτσι ήπια. Για, τις... για την τροπολογία Μπραντνερ θα ήθελα να την εξετάσω πιο προσεκτικά και να ακούσω τις εξηγήσει. Όλα αυτά πολύ συνοπτικά, μια και δεν έχω πολύ χρόνο. Ε, καλώ τους συναδέλφους να υποστηρίξουν Αυτό το προσανατολισμό που προσπαθήσαμε να σχεδιάσουμε μαζί με τον εισηγητή, τον κύριο Σαλαφράγκα. Από τους φιλελεύθερους, τρία λεπτά για την Thank Ευχαριστώ. Καταρχήν, θα ήθελα να πω ότι πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί διότι σε εθνικό επίπεδο πάρα πολλές κυβερνήσεις ε, μειώνουν τον προϋπολογισμό τους λόγω της ε, οικονομικής κρίσης. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν είναι δυνατόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο να χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερα χρήματα άρα θα πρέπει να ακολουθήσουμε την ίδια γραμμή που ακολουθούν και οι εθνικές κυβερνήσεις. Ακόμη όμως και όταν λέω κάτι τέτοιο ξέρω ότι τα χρήματα που διαθέτουμε για την ε, εξωτερική πολιτική ε, δεν είναι πολλά και είναι πολύ βασικό να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ορισμένα βασικά προβλήματα τα οποία τονίζουμε και εγώ θα ήθελα να τονίσω επιπλέον ότι η παρακολούθηση, η εποπτεία είναι <clears throat> σημαντική. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ σε τέσσερα θέματα. μου κάνει εντύπωση η αρνητική στάση του Συμβουλίου ε, σχετικά με το απόθεμα για επίγουσες περιπτώσεις ε, ε, διότι θεώρησαν ότι το τωρινό απόθεμα είναι πολύ υψηλό και έχουν μηδενίσει τις πληρωμές για το επόμενο έτος. Σύμφωνα με τους ε, διεθνείς ε, δωρητές οι οποίοι έχουν διαθέσει τα χρήματα ε, Πρέπει να πω ότι όχι μόνο η δικιά μας πολιτική ομάδα αλλά και άλλες είναι υπέρ του να διατηρήσουμε την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής των 203 εκατομμυρίων. Κάτι άλλο είναι το ε, εργαλείο σταθερότητος το, όπου θα πρέπει να αποφύγουμε τις ε, διαμάχες και θα πρέπει να έχουμε δυνατότητα να ανταποκριθούμε ε, ε, σε κρίσεις και ιδίως να συμβάλλουμε η σταθεροποίηση και στην επίλυση κρίσεων. Τρίτον, θα ήθελα να αναφερθώ στο, πρόγραμμα Ευρωπαϊκής ε, ε, Γειτονίας και πιστεύω ότι ε, υπάρχουν θέματα τα οποία απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα έπρεπε να χρηματοδοτηθούν επαρκώς διότι πρέπει να χρηματοδοτήσουμε τους ανατολικούς και νότιους γειτόνους μας οι περιοχές αυτές όντας πολύ σημαντικές και θα έπρεπε να εντείνουμε τη συνεργασία. Τέλος, το τελευταίο θέμα το οποίο θέλω να θίξω είναι η στρατηγική της Βαλτικής ε, διότι υπάρχει η ευρωπαϊκή πολιτική γυτνιάσεως και οικονομική συνεργασία με την Ανατολική Ευρώπη. Πέραν της οικονομικής πτυχής θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα για να εφαρμόσουμε την στρατηγική για τη Βαλτική. Ευχαριστώ κύριε Γιατεμάκη. Ο κύριο, η κυρία Μπραντνερ, η οποία είναι σκιώδης συγητής των Πρασίνων, έχει το λόγο για τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Θα αναφερθώ σε μερικά θέματα και στα ερωτήματα που έθεσε ο κύριος Σαλαφράγκα. Καταρχήν θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή και ευχαριστώ που είπατε ότι θέλετε να συζητήσετε τη γνωμοδότησή σας μαζί μας. Ε, σχετικά με τους αριθμούς όσον αφορά την μεσολάβηση και τη στήριξη που αναφέρατε ξέρετε ότι υπάρχει μία απόφαση του Συμβουλίου του 2009 η οποία επιζητεί μία βελτίωση της δυνατότητας ε, μεσολάβησης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αλλά δεν προβλέπεται κάποιο κονδύλι σχετικό στον προπολογισμό και ενδεχομένως δεν μπορεί να καταρτιστεί γρήγορα θα μπορούσε όμως να υπάρξει μία προκαταρτική δράση για να μπορέσει στο μέλλον να θεσμοθετηθεί. Αυτό συζήτησα και με τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επεξεργάζονται το θέμα για να δούμε ε, πώς δίκαια και χωρίς μεγάλο κόστος θα μπορέσουμε κάποια μέρα να καταλήξουμε σε μια καλή δυνατότητα διαμεσολάβησης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και πώς μπορούμε να ανοίξουμε αυτό το δρόμο και την ε, προκατατική δράση. Ε, Ευχαρίστω λοιπόν ε, θα ήθελα να κοιτάξουμε αυτό το θέμα όσον αφορά την Τινησία που είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα έπρεπε να αξιολογηθεί θα έπρεπε να έχουμε περισσότερους, περισσότερα αποθέματα και να γίνει αξιολόγηση γιατί ξέρουμε ότι δεν αποδίδει και ε, πρέπει να μπορέσουμε να ελέγξουμε πού κατευθύνεται η χρηματοδότηση αυτή. Θέλω να κάνω και ένα ερώτημα, διότι από τη μία πλευρά χαιρετίζω τις προσπάθειες του κυρίου Σαλαφράγκα να εφαρμόσει αυτά που συμφωνήσαμε με την κυρία Άστον σχετικά με τις γραμμές του προϋπολογισμού ε, του CSDP και πιστεύω ότι πάμε πολύ καλά αλλά έχουμε τη Βοσνία και άλλες περιοχές και πιστεύω ότι θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε κάποιο κονδύλι για κάθε περίπτωση και αν δεν επιτύχουμε να μπορέσουμε να τα συγχωνεύσουμε διαφορετικά θα βρεθούμε στην ίδια κατάσταση δηλαδή δεν θα μπορούμε ε, να ε, στηρίξουμε ένα χώρο χωρίς να στηρίξουμε και τους άλλους. Και η Βοσνία είναι ένα βασικό ο θέμα. Δεν αντιλαμβάνουμε λοιπόν γιατί μπορούμε να έχουμε χωριστό κονδύλι για το Αφγανιστάν και όχι για την Βοσνία. Θα πρέπει να είμαστε πιο θαραλέοι, να κατακαιρματίσουμε τα κονδύλια της εξωτερικής δράσης και ευχαρίστως να προβώ σε τροπολογίες που θα υποβληθούν στην Επιτροπή Προϋπολογισμού κατευθείαν. Όσο αναφορά τις δεσμεύσεις θα ήθελα επίσης να σχολιάσω το σημείο αυτό. Ευχαριστώ. Η κυρία μου για δύο λεπτά. Ε, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή μας τον κύριο Σαλαφράνκα και για την έκθεσή του και για την ε, ισχυρή του θέληση και για την ε, ικανότητα πειθούς που έχει. Φυσικά θέλουμε να επαναφέρουμε τα αρχικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά θα ήθελα να εκφράσω την έκπληξή μου για τροπολογίες σε συγκεκριμένες δημοσιονομικές γραμμές. Η τροπολογία 50... 28 ε, και 29.05.04. Ε, γιατί δημιουργείται μια νέα δημοσιονομική βάση χωρίς καμία δημοσιονομική γραμμή, συγγνώμη, χωρίς καμία νομική βάση. Ενώ κάθε δημοσιονομική γραμμή πρέπει να στηρίζεται σε μια νομική βάση. Ε, εδώ, αφενός ε, διασπούμε το μέσο συνεργασίας με τις βιομηχανικές χώρες αφαιρώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν ξέραμε ποιο κριτήριο από το μέσο αυτό και αφετέρου δημιουργείται μια νέα δημοσιονομική γραμμή εκτός αυτού του μέσου που είναι νεοπαγές σχετικά και δεν ξέρουμε με ποιο κριτήριο δόθηκαν σε αυτή τη νέα δημοσιονομική γραμμή 4-5 εκατομμύρια ευρώ. Ανάλογα για τώρα μιλάμε για τροπολογία Μπροκ ή για τροπολογία του σκιώδου σοσιαλιστού εισηγητού. Αυτό το μέσο συνεργασίας με τις βιομηχανικές χώρες κυρίως ε, το δικαιούνται οι Ηνωμένε Πολιτείε. Με ποιο δικαίωμα αφαιρούμε τις Ηνωμένε Πολιτείες η κατανομή των κονδυλίων γίνεται ανάλογα με τα προγράμματα που υποβάλλονται. Επίση, η τροπολογία 50.00 αφορά μόνο τα σχόλια. Δεν συμφωνώ ότι θα πρέπει να γίνει διαχωρισμό. Επίση, 50.28 και η 50.33 αφορούν επίση ε, η μία το σχό, τα σχόλια και άλλη τα σχόλια και τα ποσά και πάλι δεν ξέρω ε, ποια κριτήρια. Θα πρέπει οι πολιτικές ομάδες να επαληθεύσουν τον κατάλογο ψηφοφορίας τους, αυτή τη λίστα, γιατί ε, δεν ξέραμε ποια κριτήρια υπευλήθησαν αυτές τι τροπολογίες. Προσέξτε λοιπόν πώς θα ψηφίσετε οι πολιτικές ομάδες. Ένα άλλο θέμα, πειραματικό σχέδιο της κυρίας Γιατερμάκη για Φόρουμ Κοινωνίας των Πολιτών Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας. Έχει νόημα εν μέσω κρίσης να δημιουργήσουμε ε, να προτείνουμε πιλωτικό πρόγραμμα ενώ συστηματικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απορρίπτει τα πιλωτικά μας προγράμματα. Δεν είναι και πολύ συνεπές κάτι τέτοιο. Τέλος, ό,τι αφορά τη βοήθεια την ενίσχυση προς την Ούνρα με τον κύριο Δελβάγε προτείναμε ένα ποσό αντίστοιχο με αυτό που πραγματικά εκτελέστηκε στο προϋπολογισμό του 2009. Είναι το τελευταίο στοιχείο που έχουμε για τις ανάγκες της Ούνρα. Και στην πρόταση των εισηγητών το ποσό είναι ακόμη πιο μικρό. Γιατί? Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ την κυρία Μουνίθ. Κυρία Γκόμες, δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον εισηγητή και τους σκιώδης εισηγητές ε, για το έργο τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, να συμφωνήσω με την πρόταση για την επαναφορά του κονδυλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέσο δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και τον προϋπολογισμό για τις αποστολές παρατήρησης εκλογών. Συμφωνώ με την επαναφορά των ποσών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα κονδύλια αυτά. Επίσης θα ήθελα να υποστηρίξω την τροπολογία της κυρίας Μουνής για το 90.03.06 για τους ειδικού απεσταλμένους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ανάγκη να συμπεριληφθεί η μνήμα ότι η οι διορισμοί θα πρέπει να τηρούν ε, την ισότητα των φύλων και τις πολιτικές ισότητες φύλων. Γιατί αυτό δυστυχώς δεν ε, συνέβη μέχρι στιγμής και είναι πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να το επισημαίνει. Επίσης, ε, συμφωνώ με τις προτάσεις και τις τροπολογίες που επαναφέρουν ε, τα κονδύλια για τις αστυνομικές ε, αποστολές της ε, ΚΕΠΑ, της Κοινής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας. Νομίζω έτσι διευρύνεται και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος. Ξεχάσαμε μια εισηγήτρια, σκιώδη εισηγήτρια, η οποία όμως δεν μας είχε ζητήσει το λόγο. Ε, της δίνουμε τώρα το λόγο. Τρία λεπτά, κυρία Λόεζινγκ. Ευχαριστώ. Ε, θεώρησα ότι ούτως ή άλλως αυτομάτως θα καλέσετε όλους τους σκιώδεις εισηγητές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον κύριο Σαλαφράνκα για την ε, γνωμοδότησή του. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει σύντομα μία ρεαλιστική πρόταση σχετικά με τον ε, προϋπολογισμό που μας απασχολεί κατά τρόπον ώστε να μπορέσουμε εγκαίρως να τον ελέγξουμε και να κατανείμουμε τα διάφορα κονδύλια διότι κατά την γνώμη μας ε, ε, ήταν ε, ανεπαρκής ο χρόνος ο οποίος διετέθη ε, για την ε, παρακολούθηση αυτών των κονδυλίων διότι κατά τη γνώμη μου ε, χρειάζονται δημοκρατικές διεργασίες και διαπραγματεύσεις και τώρα κατά τον έλεγχο του προϋπολογισμού θα πρέπει να μπορέσουμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Όσον αφορά την Παλαιστίνη, η Ηνωμένη Αριστερά συμφωνεί με τον ε, κύριο Σαλαφράγκα ότι ε, δεν πρέπει να μειωθούν γιατί είναι απαραίτητα ε, τα κονδύλια αυτά για να μπορέσει να επιβιώσουν οι Παλαιστίνοι και να επιληθεί το παλαιστινιακό πρόβλημα. Ε, επίσης ε, θα πρέπει να υπάρχουν επαρκείς πόροι διαθέσιμοι σε όλα τα βασικά θέματα αλλά πρέπει να ε, είμαστε πιο ε, θετική και να προωθούμε την ειρήνη και αυτό δεν γίνεται ε, μέσω στρατιωτικών δυνάμεων. Δεν πρέπει δηλαδή να χρηματοδοτούμε στρατιωτικές επιχειρήσεις αλλά θα πρέπει ε, να ενισχύσουμε τις ειρηνικές ενέργειες όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διαμεσολαβητική και όχι ε, παράγων που επιτίθεται και αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στις διάφορες γραμμές του προϋπολογισμού. Συμφωνούμε ότι εάν υπάρχει ε, βοήθεια προς τους πολίτες αποκλειστικά θα πρέπει να προωθείται κατά προτεραιότητα. Ευχαριστώ κύριε Λέζινγκ. Μίλλερ από τη Γενική Διεύθυνση Ραγλέξης Κομισιόν. Αν μπορείτε, όχι πάνω από πέντε λεφτά, σας παρακαλώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο, Πρόεδρε. Καταρχάς, όπως είπαν πολλοί βουλευτές, ε, καταλαβαίνουμε ότι η οικονομική κατάσταση είναι δύσκολη. Αυτό είναι το δύσκολο πλαίσιο της στο οποίο ζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και καταλαβαίνω ότι Πολλοί βουλευτές ζητάνε να είμαστε αυστηροί και λυτοί. Συμφωνούμε. Ε, θα ήθελα να πω επίσημα ότι χαιρόμαστε φέτος για την υποστήριξη της Επιτροπής και του κ. Σαλαφράγκα ε, για την επαναφορά των αρχικών κονδυλίων της Κομισιόν που, επί των οποίων πρότεινε ε, περικοπές, κυρίως για τα διοικητικά θέματα διοικητικά έξοδα, αλλά και κυρίω όλα τα μέσα του τίτλου 4 και κυρίω το πρωταξιακό μέσο. Ο κ. Σαλαφράγκα δεν επαναφέρει τι προτάσει μα για το μέσο αναπτυξιακή συνεργασία και το μέσο γειτονία. Δύο μεγάλα μέσα. Καταλαβαίνουμε από την άλλη τις προσπάθειες που κάνει ο κ. Σαλαφράγκα, αλλά οποιαδήποτε μείωση στην διοικητική υποστήριξη αυτών των μέσων μπορεί να μας δημιουργήσουν προβλήματα για την υλοποίηση το, την εφαρμογή κατά 100% του προπολογισμού. Το θέμα της Παλαιστίνης επίσης ετέθη από πολλούς βουλευτές. Σημειώνουμε την πρόταση αύξηση της γραμμής του προλογισμού κατά 100 εκατομμύρια από 200 σε 300 εκατομμύρια που θα το επαναφέρει στα επίπεδα που είχε αρχικά προτείνει η Κομισιόν σε προηγούμενους ε, προϋπολογισμούς. Αυτό που θα ήθελα να πω για αυτό το σημείο είναι ότι η κυρία Άστον και η Κομισιόν θα ήθελα να υπάρχει υποστήριξη προς, την, προς τον παστινιακό λαό και να μην μειωθεί σε σχέση με τα προηγούμενα δύο-τρία χρόνια. Μία από τις περικοπές που προτείνει ο κύριος Σαλαφράγκα που σε σχέση με την πρόταση του Αφγανιστάν σε σχέση με την πρόταση συγγνώμη, ε, της Κομισιόν για το Αφγανιστάν προγραμματίζουμε τη βοήθειά μας σε χώρες όπως το Αφγανιστάν πολύ προσεκτικά. Ε, ο προγραμματισμός συζητείται με όλους τους εμπλεκόμενους, τους εταίρους, ε, τα κράτη-μέλη και το Κοινοβούλιο. Οποιαδήποτε περικοπή σε αυτή τη γραμμή του προπολογισμού θα ήταν περικοπή στη βοήθειά μας υπέρ του αφγανικού λαού. Θα ήθελα τώρα να πάω στην ΚΕΠΑ. Υπάρχουν ε, δύο διαστάσεις στην ε, τροπολογία. Καταρχάς είναι η διαφάνεια και δεύτερον είναι ένα αποθεματικό που με την υποστήριξη των ε, συσιαλιστών ο κ. Σαλαφράγκα θέλει να δημιουργήσει για τις γραμμές κατεπίγουσας βοήθειας. Ο κ. Σαλαφράγκα θέλει να υπάρχει διαφάνεια για την ΚΕΠΑ και νομίζω ότι αυτή η προσπάθεια λαμβάνεται υπόψη πολύ σοβαρά. Αλλά για να επιτύχουμε τη διαφάνεια πρέπει να δημιουργήσουμε ξεχωριστές γραμμές προϋπολογισμού για κάθε αποστολή της ΚΕΠΑ. Γιατί αυτό που προτείνει ε, η Επιτροπή είναι 8 διαφορετικές γραμμές για 8 διαφορετικές αποστολές. Δεν νομίζουμε ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να επιτύχουμε τη διαφάνεια αυτός. Ήδη δίνουμε λεπτομερείς πληροφορίες για τον προϋπολογισμό της κάθε αποστολής, δίνουμε αυτά στοιχεία στην Επιτροπή και πριν από κάθε αποστολή, ή μάλλον μετά από την υιοθέτηση κάθε αποστολή από το Συμβούλιο, μέσα σε πέντε μέρε σα στέλνουμε επίση και το λεπτομερή προπολογισμό τη ε, συγκεκριμένη αποστολή. Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε λοιπόν αυτό το θέμα με το Κοινοβούλιο και να βρούμε άλλους τρόπους για να εξασφαλίσουμε την διαφάνεια. Οτιδήποτε συμφωνηθεί στο κεφάλαιο της ΚΕΠΑ θα πρέπει να συμφωνηθεί επίσης και με τα κράτη-μέλη ε, και το Συμβούλιο ε, στα πλαίσια της διαδικασίας ε, προϋπολογισμού. Επίσης, με αυτό το πνεύμα καταλαβαίνουμε και τη δημιουργία του αποθεματικού. Ε, νομίζουμε ότι είναι μια βάση ούτω ώστε το Κοινοβούλιο πάνω σε αυτή θα μπορούσε αργότερα στα πλαίσια της διαδικασία προϋπολογισμού να, να συζητήσει με το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη. Αλλά το αν θα διατηρηθεί αυτό το αποθεματικό στον προπολογισμό αν διατηρηθεί συγγνώμη, το αποθεματικό αυτό ε, στον προπολογισμό τα επόμενα χρόνια, μπορούμε να, μπορεί να μειώσουμε την δυνατότητα απόκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κρίσεις κτλ. Τέλος, για την ΕΑΣ, την Υπηρεσία, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, ο Κρίστοφερσον, ο κ. Κρίστοφερσον, εκπρόσωπο τη κυρία Άστον, είναι μέσα στην αίθουσα και μπορεί και αυτό αργότερα να πάρει το λόγο και να σα επιβεβαιώσει αυτά που θα σα πω. Καταλαβαίνουμε οπωσδήποτε την ανάγκη που εξέφρασαν πολλοί βουλευτέ να γνωρίζουν τι γίνεται με τον προπολογισμό αυτό τη εξωτερική υπηρεσία το συντομότερο δυνατόν. Και η Κομισιόν ετοιμάζει μια τροπολογία αυτή τη στιγμή του προπολογισμού. Αυτή τη στιγμή προετοιμάζεται. Ε, όταν βγω από αυτήν την αίθουσα θα πω και εγώ να ασχοληθώ με αυτό το θέμα. Θέλουμε με αυτή την πρόταση να υιοθετηθεί, αυτή η πρόταση να υιοθετηθεί από το Συμβούλιο στις 15 ε, Σεπτεμβρίου. Είναι τροποποιητική επιστολή και η συνθήκη μας επιτρέπει μέχρι την πρώτη ανάγνωση στο Κοινοβούλιο να παρουσιάσουμε μια τέτοια τροποποιητική επιστολή. Ε, θα είμαστε έτοιμοι λοιπόν για την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου με αυτή την επιστολή. Αυτή τη στιγμή η κυρία Άστον ε, εμπλέκεται στην προετοιμασία αυτής της απόφασης, η οποία τρέχει ακόμα. Ευχαριστώ λοιπόν ακόμα μια φορά τον εισηγητή για την ε, προθυμία να συνεργαστεί μαζί μας, να ακούσει τις ανησυχίες μας και ελπίζουμε να συνεχίσουμε αυτή την ε, εποφελή συνεργασία με την Επιτροπή σας τις επόμενες φάσεις της διαδικασίας. Ευχαριστώ. Τελικά σχόλια θα τα κάνει τώρα ο εισηγητής, ο κ. Σαλαφράγκα. Ευχαριστώ. Ακούσαμε όλους ε, τους συναδέλφους σχεδόν και θα ήθελα να απαντήσω ατομικά στον, καθ, καθένα. Ευχαριστώ κύριε Γουαλτιέρη για αυτά που είπατε. Μείνετε ήσυχος για την Παλαιστίνη γιατί η Σύσσωμη Επιτροπή στηρίζει το αίτημα ενίσχυση τη Παλαιστινιακής Αρχή. Και γνωρίζουμε κάλλιστα τι λεπτομέρειε τη Συμφωνία της Μαδρίτης ό,τι αφορά την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερική δράση. Και συμμερίζομαι τις ανησυχίες σα ε, για το κατά πόσο είναι βιώσιμο δημοσιονομικά το αίτημα ειδικού απεσταλμένου για το Θιβέτ. Υπάρχουν πολλές αντεδείξει από άποψη διπλωματικής πρακτικής για την πρόβλεψη μιας τέτοια θέση ενό τέτοιου αξιώματο. Τώρα, για το θέμα τη Τινησία, το... σίγουρα οι πράσινοι έχουν πρόβλημα, αλλά εγώ δεν ήθελα μέσω σχολείων να, να στιγματίσουμε οποιαδήποτε χώρα, γιατί υπάρχουν και άλλα μέσα πέραν του προπολογισμού για να εξασφαλιστεί αποτελεσματικό έλεγχο σε ό,τι αφορά την ε, συνεργασία, σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα Εθνικής Συνεργασίας με την Τινησία. Έγινε και με άλλες χώρες της περιοχής, ε, αλλά και όχι μόνο αυτής της περιοχής και με άλλες χώρες του πλανήτη. Και δεν νομίζω ότι ε, είναι σκόπιμο με ένα σχόλιο στον προπολογισμό να προσπαθούμε να λύσουμε ένα τέτοιο ζήτημα. Ευχαριστώ την κυρία Γιατεμάκη για τα σχόλιά της. Εμένα δεν με κατέπληξε η αρνητική θέση του Συμβουλίου, γιατί στην δημοσιονομική συζήτηση Έχουμε καταρχήν μία πρόταση που είναι φάρος κατά κάποιο τρόπο και κατόπιν γίνονται διάφορες διαπραγματεύσεις, διελκυστίνδες και προχωρούμε σε μια δημοσιονομική διαδικασία που έχει και μια κατάληξη. Αυτά σε ό,τι αφορά κύριε για την μάκη τις επιχειρησιακές γραμμές νομίζω ότι είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι από τη λύση. Εγώ είμαι διαλλακτικός και ελπίζω και άλλοι συνάδελφοι να δούμε το θέμα των πιστώσεων πληρωμών, γιατί οι πιστώσεις πληρωμών σηματοδοτούν τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης ό,τι αφορά την ικανοποίηση των ε, κρεμουσών της ε, υποχρεώσεων. Σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες και το θέμα της συνοχής ε, το συζητήσαμε τώρα για τις πιστώσεις πληρωμών θα επιληφθώ του θέματος για να δω αν μπορούμε να ικανοποιήσουμε ακόμη περισσότερο την κυρία Γιατενμάκη. Πάντως, αντιλαμβάνομαι και την ανησυχία σας για την ΑΕΤ και τη συμμερίζομαι. Και κάτι άλλο που ξέχασα στην εισαγωγή είναι το θέμα της βοήθειας προς το Πακιστάν. Αλλά αυτό το θέμα άφεται περισσότερο των αρμοδιοτήτων ε, της Επιτροπής Ανάπτυξης. Δεν θα πρέπει να μπαίνουμε στα χωράφια τους, γιατί υπάρχει μια κατανομή των αρμοδιοτήτων και θα πρέπει να την ε, σεβαστούμε. Ούτε γνωρίζουμε τι θα γίνει με τα 70 εκατομμύρια για το προϋπολογισμό του 2011 που ήδη έχουν προβλεφθεί για τις ανάγκες του Πακιστάν. Κυρία Μπράντνερ, εγώ θεωρώ ότι οι όροι της συμφωνίας του Συμβουλίου και εδώ απαντώ και στις ανησυχίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπουν μόνο μερικές έκτακτες αποστολές να αναφερθούν ε, ατομικά. Σε ό,τι αφορά όμω την ε, δημοσιονομική διαφάνεια, καλύτερα να μην γίνει η λεπτομεριακή κατανομή απαρίθμηση των συγκεκριμένων αποστολών. Σε ό,τι αφορά τα πιλωτικά προγράμματα, συμφωνώ με την πρόταση του πιλωτικού προγράμματο, αλλά ε, με μειωμένο ποσό σε σχέση με αυτό που προτείνει η κυρία Μπράντνερ. Κυρία Μουνή, σε ό,τι αφορά τη διμερή συνεργασία με τις ε, Ηνωμένε Πολιτείε. Η δράση αυτή είναι συμπληρωματική δράση, επουδενή δεν ε, περιορίζει τη, τα κονδύλια για τη συνεργασία με τις βιομηχανικές εκβιομηχανισμένες χώρες. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διευκρινίζει αν γίνεται ταξινόμηση με βάση τις ετήσιες ε, υποχρεώσεις, αλλά θα ήθελα να σας επισημάνω ότι στο τελευταίο ψήφισμα που εγκρίναμε για τις διατελαντικές σχέσεις ζητήσαμε η δημοσιονομική προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μελέτες ή δραστηριότητε που ευνοούν τις ε, διατελαντικές σχέσεις θα πρέπει να την υπόψη όχι μόνο τα think tanks που κατοικοδρεύουν στι ΗΠΑ, αλλά χωρί επαναλαμβάνω, να ε, παραβιάσουμε τις δεσμεύσει μας με τις ΗΠΑ, να δώσουμε περισσότερη έμφαση σε οργανισμούς και think tanks ε, που εδρεύουν στην Ευρώπη και έχουν και ευρωπαϊκή συνιστόσα. Τώρα, με βάση τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με μια μικρή αύξηση και με την πολιτική υποστήριξη των ψηφισμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κρίναμε σκόπιμο να βρούμε μια συμβαστική λύση στην ε, τροπολογία Μπροκ. Επαναλαμβάνω, αυτό θα γίνει ει βάρο των ποσών που προβλέπεται για τη συνεργασία με τι εκβιομηχανισμένε χώρε. Πρόκειται για συμπληρωματικά ποσά. Επίση, ευχαριστώ την κυρία Γκόμε για τα σχόλιά τη και την μεγάλη τη ευαισθησία για τα ζητήματα ασφάλεια και τη υποστήριξη των αποστολών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλος, ε, κυρία Λέσινγκ, χαίρομαι που συμφωνείτε όπως ε, ευτυχώς μας είπε και ο πρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα της παρουσίασης του προϋπολογισμού από τις 15 Σεπτεμβρίου για την ΕΑΣ. Συμφωνώ επίσης με τα ποσά που προτείνουμε για την Παλαιστίνη. Κατέγραψα τις ανησυχίες του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις διοικητικές δαπάνες, ιδιαίτερα για την πολιτική γειτονία. Μέχρι τη Δευτέρα θα συνεννοηθώ με τους συναδέλφους για να δούμε αν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Και επίσης ε, η δημοσιονομική διαδικασία γνωρίζεται ότι είναι και θέμα τακτικής. Και η θέση μας στην συνεδρίαση της Δευτέρας θα τύχουν περαιτέρω διαπραγμάτευση και με την Επιτροπή Προπολογισμών που θα εγκρίνει και τις τροπολογίε. Ήδη ξεπεράσαμε το όριο του αποθεματικού με τα 18 εκατομμύρια που προτείναμε. Θα γίνουν διάφορες προσαρμογέ και ελπίζω να διασκεδαστεί και η ανησυχία του κυρίου Γουαλτιέρη ότι θα συνταχτούμε όλοι με μια σαφή θέση της Επιτροπής μας για τις προτεραιότητές μας ώστε κατά την περάτωση της δημοσιονομικής διαδικασίας οι δικές μας προτεραιότητες να μην ε, αλλοιωθούν στο πλαίσιο της τελικής απόφασης που θα λάβει η Επιτροπή Προϋπολογισμών. Θα προσπαθήσω πάντως, επαναλαμβάνω, να λάβω υπόψη τις ανησυχίες σας και να βελτιώσω την έκθεση με τη γενική θέση της Επιτροπής μας. Αυτά και ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους για τη συμμετοχή και τη συνεργασία τους. Ευχαριστώ και εγώ τους συναδέλφους, προφανώς τους ε, εισηγητές. Η ψηφοφορία θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής ή μάλλον στην επόμενη Ολομέλεια στις 6 Σεπτεμβρίου. Πάμε στον χρηματοδοτικό κανονισμό και στις τροπολογίες αυτού. Απαραίτητες αλλαγές, ούτως ώστε να μας επιτρέψουν να να επιτρέψουν στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης να λειτουργήσει σωστά. Όπως ξέρετε, σε αυτή τη φάση η τροπολογία του δημοσιονομικού κανονισμού συνδέεται με το καθεστώς και το κανονισμό για τους δημοσίους υπαλλήλους. Ο Σάριος Βόλσκι την επόμενη Δευτέρα θα παρουσιάσει την έκθεσή του για την τροπολογία του καταστατικού. Και σήμερα έχουμε την ε, ενδιαφέρουσα αυτή έκθεση του συναδέλφου φάρ για τον προϋπολογισμό αυτό. Ο, οι κύριοι Μπροκ και οι ο κύριος Φερχόφσταντ συνεργάστηκαν μεταξύ τους και με τον κύριο Γκουαλτιέρη το κέντρο βάρους της, δημοσιο... της ε, νομοθετικής διαδικασίας μετατίθεται τώρα. Η νομική υπηρεσία για το καθεστώς των ε, υπαλλήλων και η Επιτροπή Προϋπολογισμών και Ελέγχου του Προϋπολογισμού για το προϋπολογισμό φυσικά της ΕΑΣ είναι απόλυτα υπεύθυνη, ενώ εμείς προφανώς ως, ε, έκθεση, ως ε, Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ε, ασχολούμαστε και εμείς με, αυτή την, αυτό το σημείο. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Κύριε Φάρμ, όσο μπορείτε πιο γρήγορα, αν γίνεται μέσα σε 5-6 λεπτά, να μας παρουσιάσετε την έκθεση αυτή. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομος ε, γίνεται. Όπως είπατε ε, αυτή είναι η συμβολή μας στην αλλαγή του δημοσιονομικού καλογινισμού λόγω της ε, υπηρεσίας εξωτερικής δράσεως και εδώ μπορούμε όντως να επηρεάσουμε την κατάσταση. Η βάση για τη γνωμοδότηση αυτή είναι η συμφωνία της Μαδρίτης για την υπηρεσία ευρωπαϊκής εξωτερικής δράσεως και διατυπώσαμε ε, τροπολογίες για να μπορέσει να συνάδει ο κανονισμός με ό,τι ελέγχθη στη Μαδρίτη. Υπάρχουν όμως τομείς που δεν έχουν καλυφθεί από τη Συμφωνία της Μαδρίτης ή που είναι πιο γενικά θέματα που θέλουν καλύτερα ρύθμιση. Γι' αυτό και εξετάσαμε πιο ενδελεχώς το θέμα ε, ιδίως ε, λαμβάνοντας υπόψη την ιστορική προοπτική ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προσφορά ειρήνης και την προσαρμογή εις το νομοθετικό έγγραφο. Είναι πιο βασικός ο σχολιασμός των τροπολογιών, των τροπολογιών 7, 8 και 9. Στο 7 ζητούμε η υπηρεσία εξωτερικής δράσης να θεωρηθεί σαν ένα θεσμικό όργανο το οποίο ε, θα πρέπει να προβλέπει και ε, κάποιον υπολογισμό χρηματοδότησης και δαπανών όπως και στις ε, άλλες υπηρεσίες και επίσης αναφέρουμε μόνο δύο από τις, τους τρεις επιτρόπους που εμπλέκονται και θα έπρεπε να αναφερθούμε και στην κυρία Γιώργεβα σε αυτά τα συμφραζόμενα είναι κάτι που θα εξετάσουμε. Τώρα, το πιο βασικό είναι το σημείο όπου ζητούμε ένα έγγραφο εργασίας το οποίο να παρουσιάζει συνολικά τον προϋπολογισμό. Όλα τα διοικητικά και επιχειρησιακά έξοδα και λεπτομερώς απαριθμούμε πώς το έγγραφο αυτό πρέπει να παρουσιάζεται. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να γίνει σωστά. Στην τροπολογία 9 ε, υπησερχόμεθα σε περισσότερες λεπτομέρειες από ό,τι είχε προβλέψει η Συμφωνία της ε, Μαδρίτης όσον αφορά την ηγεσία και τον υπεύθυνο διαχειριστή, ποιος δηλαδή ευθύνεται κτλ. Αυτές είναι οι πιο βασικές τροπολογίες αλλά υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν έχω ακόμη περιλάβει και θα έπρεπε να συζητήσουμε στην Επιτροπή τι θέλουμε να πράξουμε. Καταρχήν όσον αφορά τον προπολογισμό του 2011 και τις γραμμές του προπολογισμού που μας ενδιαφέρουν για τις αποστολές διότι ε, όπως ξέρετε ε, είναι ένα θέμα το οποίο ε, έχει προβλεφθεί στην ημερήσια διάταξη αναφέρεται στη διαθεσμική Συμφωνία αλλά αναφέρεται στην εποχή πρώτης συνθήκης της Λισαβόνας και πρέπει να δούμε τώρα πώς πρέπει να κατακαιρματίζεται και να παρουσιάζεται ο προπολογισμό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχω μία ιδέα προς την οποία θα μπορούσα να δεχτώ αυτό. Δηλαδή ότι αυτό δεν θα πρέπει να προβλεφθεί στη διαθεσμική συμφωνία αλλά στο δημοσιονομικό κανονισμό. Οπότε θα μπορέσουμε να περιλάβουμε μία τροπολογία στη γνωμοδότηση αυτή η οποία θα πραγματεύεται την συζήτηση που μόλις κάναμε σχετικά με τις γραμμές του προπολογισμού που αναφέρονται στην ε, την πολιτική αυτή. Επίσης ε, ένα άλλο θέμα το οποίο έχουν θίξει οι μέλη της Επιτροπής είναι ότι για να γνωρίζουμε όλα τα στοιχεία των δαπανών δεν επαρκεί να ξέρουμε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά ποιες είναι και οι συνδρομές των κρατών μελών στην πολιτική αυτή διότι διαφορετικά δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε εμείς δεν θέλω να παρέμβω με την κατανομή δυνάμεων μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κρατών μελών, αλλά νομίζω ότι είναι ένα θέμα βασικό. Αυτά είναι τα πιο βασικά στοιχεία και έχω και μερικά σχόλια ε, για σημεία όπου θα έπρεπε να κάνουμε κάποια προσθήκη και ορισμένες τεχνικές αλλαγές ε, και ε, όπου χρειάζονται τροπολογίες πριν από την επόμενη εβδομάδα. Καταρχήν να ρωτήσουμε αν ε, πρέπει να υποβάλουμε μία τροπολογία σχετικά με αυτές τις εξωτερικές αποστολές και, το ούτω καθεξής. Ευχαριστώ κύριε Φάρμ για τη δουλειά σας, για την παρουσίασή σας και για το σεβασμό του χρόνου. Μπροκ, τρία λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να κάνω μια σύντομη παρατήρηση. Ευχαριστώ τους συναδέλφους και τον συνάδελφο και πιστεύω ότι είναι στο σωστό δρόμο και μπορούμε να στηρίξουμε τις τροπολογίες που έχει υποβάλει διότι είναι στα πλαίσια της συμφωνίας όσον αφορά τη διαφοροποίηση όσον σχετικά με την παρουσίαση νομίζω ότι υπάρχει δήλωση της υπάτου ε, ε, του επιτετραμένης για το, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το κατά πόσο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα στοιχεία διότι εδώ πρέπει να καλυφθεί και ε, το μέλημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για διαφάνεια συνδεδιασμένη με ε, ευελιξία και πρέπει να βρούμε ε, μία συμβιβαστική λύση όπως το είχε πει και ο κύριος Γκουαλτιέρη. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας παρακαλέσω ώστε δυνατόν πιο γρήγορα να συζητήσουμε εδώ τον κανονισμό προσωπικού γιατί πολλά πράγματα αλλάζουν και θα πρέπει να σεβαστούμε το χρονοδιάγραμμα. Έχουμε χάσει πάρα πολύ ε, χρόνο ε, λόγω της ε, καθυστερημένης εφαρμογής των συνθηκών και ούτω καθεξής και τώρα βλέποντας πώς εκπροσωπείται η Ευρώπη στη Washington στις συζητήσεις για τη Μέση Ανατολή και ούτω καθεξής νομίζω ότι έφτασε η ώρα να έχουμε μία αρμόδια υπηρεσία, να μην υποφέρει η ποιότητα των υπηρεσιών και δεν χρειάζεται να χάνουμε, να δημιουργούμε επιπλέον χρονικά προσκόμματα. Λοιπόν, νομίζω ότι σκόπιμο θα ήταν να διεκπαιρεώσουμε αυτή την δημοσιονομική γνωμοδότηση, να συζητήσουμε μιλήσουμε και για τον προπολογισμό, να δούμε τι γίνεται με την νομική υπηρεσία, να δούμε πώς προχωρούμε, διότι θέλουμε να έχουμε μία αποτελεσματική εξωτερική περιοχή και ε, ε, ε, επιτροπή και ίσως η νομική επιτροπή και η επιτροπή προπολογισμού έχουν διαφορετικές προτεραιότητες και δεν χρειάζεται πάντοτε εμείς να προσαρμοζόμαστε. Εμείς πρέπει να εξασφαλίζουμε τα δικά μας συμφέροντα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μπραντνερ, Κυρία Μπραντνερ, για τρία λεπτά. Συγχαίρω τον κύριο Φάρμα για τη γνωμοδότηση, γιατί υπάρχουν και κάποια σημεία που αφορούν όλος ιδιαίτερος την ΑΦΕΤ, όπως είπε και ο κύριος Μπροκ. Για το άρθρο 10 έχω μια ερώτηση. Για τους ε, επικεφαλής των αποστολών ε, και την, το γεγονός ότι ότι δεν έχουμε αρμοδιότητες, δεν έχουν αρμοδιότητες μάλλον οι αντιπροσωπείες. Ε, Δεν θα πρέπει νομίζω η Κομισιόν να έχει την εξουσία να αλλάζει τα οικονομικά στοιχεία για τις αποστολές αυτές. Θέλω μια διευκρίνηση για αυτό το σημείο. Μ' αρέσει η τροπολογία 12. Ε, να είναι υπόλογοι οι εθνικοί διπλωμάτες. Ευχαριστώ, κύριος Γκουαλτιέρη, για τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φάρμα μας παρουσίασε το κείμενό του, που είναι θετικό και χρήσιμο. Δεν θα επανέλθω σε αυτά που είπε, γιατί τα συμμερίζομαι απόλυτα. Θα ήθελα να τονίσω ότι πολιτικός πώς ε, το κείμενο αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο με τα πράγματα που λέει, αλλά και με τα πράγματα που δεν λέει. Σε σχέση με το κείμενο της εισηγήτρια της Επιτροπής Προπολογισμού, ιδίω το άρθρο 1 του Δημοσιονομικού Κανονισμού, την ε, απαρίθμηση δηλαδή των ε, θεσμικών οργάνων. Η δομή που προτείνει, ε, στην οποία εντάσσει και την ΕΑΣ μαζί με το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που αντιμετωπίζονται ως θεσμικά όργανα. Δηλαδή, έχει νόημα να αντιμετωπίσουμε το Συμβούλιο ως θεσμικό όργανο. Οι πολιτικές ομάδες με το να μην παρουσιάσουμε τροπολογία δίνουμε ε, ένα μήνυμα, στέλνουμε ένα μήνυμα ότι δεν θέλουμε να αρχίσουμε μια συζήτηση για την ε, ε, για τον επαναπροσδιορισμό των θετικών θεσμικών οργάνων, αλλά κυρίω για το, τη νέα στην ε, υπηρεσία εξωτερική δράση. Για τα υπόλοιπα σημεία συμφωνούμε με τον κύριο Φάρν. Μπορούμε να βελτιώσουμε μάλιστα την πρόταση. Τώρα, αν στον δημοσιονομικό κανονισμό θα βάλουμε αναφορές στην ε, νέα δομή του προϋπολογισμού της Αλίας, εδώ με αυτόν τον τρόπο δεν θα πρέπει να αλλάζουμε τον αριθμό των γραμμών, αλλά θα πρέπει να πούμε, να κάνουμε μία αναφορά ε, αναφοράς. Η διαδικασία προϋπολογισμού καθορίζει πόσες γραμμές ή μάλλον πόσες ε, αποστολές θα έχουν δική τους γραμμή προϋπολογισμού, αν θέλετε. Και με αυτόν τον τρόπο δεν νομίζω ότι θέτουμε να αμφιβόλο την ευελιξία του προϋπολογισμού της ε, αλίας. Όλα τα ποσά μπορούν να μπουν στο εσωτερικό ενός, ε, ενός τίτλου ε, χωρίς να έχουμε απίστευτα δύσκολες και μακροσκελείς διαδικασίες. Ευχαριστώ. Ο κ. Κρίστοφσεν, εκ, εκπρόσωπος της ε, είπα της εκπροσώπου και αντιπροέδρου κ. Σάστον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που είπατε ότι η Επιτροπή ΑΦΕΤ θα παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυ στο θέμα αυτό. Νομίζω ότι είναι καλό για όλους αυτή η προσοχή που δίνεται. Ευχαριστώ τον κύριο Φάρμα για την ε, έκθεσή του, για το σχέδιο εκνομοδότησής του δηλαδή. Σωστά είπε ότι είμαστε στον τομέα της συναπόφασης εδώ. Παρότι επίσημα όταν αποφασίσαμε τον Ιούλιο τα βασικά στοιχεία δεν ήμασταν επίσημα ε, στα πλαίσια τη διαδικασίας ε, της συναπόφασης. Παρ' όλα αυτά λειτουργούσαμε σαν να είμαστε. Και το κείμενο που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο είναι ακριβώς το ίδιο με τη γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου. Το κείμενο του Συμβουλίου λοιπόν της 6 Ιουλίου προσωμιάζει στο κείμενο του Κοινοβουλίου. Γι' αυτό είναι και σημαντική η συμφωνία της δεύτερης φάσης του, του Ιουλίου. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι το κείμενο σέβεται ακριβώς αυτή τη συμφωνία του Ιουλίου. Το κείμενό σας. Δεν έχω καμία δυσκολία με το κείμενο. Σωστά είπε ο κ. Φάρμ ότι η τροπολογία 8 είναι σημαντική, λεπτομερής. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τέτοιες πληροφορίες. Με πληροφορίες όπως μας τη ζητάτε στην τροπολογία αυτή. Για τα πιο τεχνικά στοιχεία, για το πώς θα διατυπώσουμε τα σημεία, αυτά μπορούμε να, το, αυτά μπορούμε να τα δούμε στα πλαίσια κάποιων επαφών που θα είχαμε. Πάντω να μην ξεχάσουμε αυτό που εννοούσε αρχικά το 8-5. Πρέπει να υπάρχει μια επισκόπηση του τι κάνει όχι μόνο η ΕΑΣ, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση στις τρίτες χώρες. Όχι μόνο η ΕΑΣ, αλλά και η Κομισιόν. Δεν είναι λειτουργικά, είναι και διοικητικά τα έξοδα. Γιατί όταν δείτε τι λεπτομέρειες, οι λεπτομέρειε αυτές μιλάνε αποκλειστικά και μόνο για τα διοικητικά έξοδα. Για τα σχόλια του κ. Φέρν τώρα. Για το αν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία που μας δίνει ο δημοσιονομικός κανονισμός για να μεταφράσουμε το πολιτικό σημείο της πολιτικής δήλωσης σε έργο, σε πράξη. Αυτό δεν είναι κάτι που μπορώ να κρίνω εγώ. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι έμεσα αναφερόταν στην δήλωση για την πολιτική λογοδοσία ότι αυτό το πρόβλημα θα τεθεί στα πλαίσια της ευρύτερης διοργανικής συμφωνίας. Μια και νομίζω ότι όλοι θέλουν τα θεσμικά όργανα να σεβαστούν αυτό που συμφωνήθηκε τον Ιούλιο. Κυρία Μπράντερ, ποια είναι η ερμηνεία μου για το δικαίωμα απόσυρσης. για τους επιμέρους επικεφαλής των αντιπροσωπιών. Θα σας το δώσω αυτό κάποια άλλη στιγμή. Ευχαριστώ κύριε Κρίστοφερσον. Αφήνουμε τον κύριο Φεύ να μας κάνει τα τελικά συμπεράσματα, τις τελικές παρατηρήσεις και να σχολιάσει τη θέση της Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Φέρμα. Ε, Ευχαριστώ για τα σχόλια. Από ό,τι βλέπω συμφωνούμε ως προς τη γνωμοδότηση. Έχω να σχολιάσω δύο πράγματα. Καταρχήν προς την κυρία Μπράντνερ. Συμφωνώ καταρχήν με τον κύριο Κριστόφερσον ότι εδώ μιλούμε για συγκεκριμένες καταστάσεις, εξατομικευμένες καταστάσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να αλλάξει την αρχή το ρόλο, αλλά το εφαρμόζει μεμονωμένα. Ως προς αυτό συμφωνούμε. μιλήσαμε για την παρουσίαση των δημοσιονομικών γραμμών της ΚΕΠΑ. Μέχρι στιγμής είχαμε τη διοργανική συμφωνία που θα πρέπει να μεταφραστεί σε δημοσιονομικό κανονισμό. Θα πρέπει να το ξανακοιτάξουμε αυτό, να κοιτάξουμε το σαφές περιεχόμενο της διοργανικής συμφωνίας. Δεν ξέρω αν η μεμονωμένη παρουσίαση των δημοσιονομικών γραμμών είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να φανταστούμε για τη διοργανική συμφωνία ή προτιμούμε το δημοσιονομικό κανονισμό. Θα πρέπει... Νομίζω ότι η συμφωνία της Μαδρίτης αποκλείει τη δική μου πρόταση, αν και εγώ το ερμηνεύω διαφορετικά, αλλά στο ξαναελέγξουμε. Το σημαντικό είναι να βρεθεί λύση. Γιατί πάνε πάνω από 10 χρόνια που συζητούμε για το πώ θα πρέπει να παρουσιαστεί ο προπολογισμό τη ΚΕΠΑ. Είμαι ανοιχτό στι λύσει. Εγώ πάντως προτιμώ χωριστό δημοσιονομικό κανονισμό γι' αυτό παρά τη διοργανική συμφωνία. Ε, Ευχαριστώ κύριε Φέρμ. Μια ενημέρωση τώρα για το χρονοδιάγραμμα. Ο χρόνος για την παρουσίαση των τροπολογιών είναι η 7η Σεπτεμβρίου μέχρι τις 6 ε, το απόγευμα. Δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι για λόγους επικαλύψεων με άλλες ψηφοφορίες στην Επιτροπή Προϋπολογισμού, Προϋπολογισμών και Ελέγχου του Προϋπολογισμού και λόγω της πίεσης του χρόνου. Ζητώ συγγνώμη από όλους όσους δεν έχουν μετρική γλώσσα τα αγγλικά, όπως εγώ εξάλλου, αλλά οι τροπολογίες θα καταδεθούν αναγκαστικά μόνο στα αγγλικά. 20 Σεπτεμβρίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή και Εκτιμούμε ότι τη δεύτερη σύνοδο Ολομέλειας του Οκτωβρίου θα ψηφίσουμε. Τώρα, για τις επόμενες συνεδριάσεις. Στις 6 Σεπτεμβρίου, από στις 7 η ώρα το απόγευμα, θα συνεδριάσουμε και στις 7 Σεπτεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, θα συνεδριάσουμε επίσης αυτές είναι οι επόμενες συνεδριάσεις μας. Γεια σας.